Possiamo dare inizio a questa importante commissione straordinaria. Παρακαλώ πολύ καθίστε να ξεκινήσει αυτή η έκτακτη συνεδρίαση. Per favore prendete tutti posto, diamo inizio. Παρακαλώ πολύ καθίστε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ο Πρόεδρος παρακαλεί να καθίσουν όλοι εν ηρεμία για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Bene, cari Καλωσορίσατε αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίσατε όλοι οι συνάδελφοι του συναδέλφου. Ε, καλώς ήρθατε και στην Κομισιόν και στην ε, Ιρλανδική Προεδρία, στη διαπραγματευτική ομάδα σε όλους. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι η διαπραγματευτική ομάδα στην τελευταία από τους περίπου 40 τριμερείς διαλόγους ε, που απασχόλησαν την Προεδρία, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν ότι επετεύχθη μια πολιτική συμφωνία επί των τεσσάρων φακέλων ε, περί των οποίων γίνεται λόγος. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για πολιτική συμφωνία. Υπενθυμίζω επίσης ότι σήμερα δεν θα ψηφίσουμε. Βεβαίως θα ακολουθήσουμε την συνήθη διαδικασία ψηφοφορίας αφού θα έχουν αναλυθεί όλα τα νομοθετικά κείμενα και αφού φυσικά θα έχει υπάρξει συμφωνία όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως θα αναλύσουμε την έκβαση αυτής της συμφωνίας και επομένως μετά τις παρουσιάσεις των εκδιεξιών μου καθημένων ε, συναδέλφων κάμπος για άμεσες επιδοτήσεις Μισελ Νταντέν, Καπούλα Σάντος όσον αφορά το θέμα για την εποπτεία της ΚΑΠ ε, και μετά λοιπόν από την παρουσία των πολιτικών συμφωνιών από την πλευρά των εισηγητών θα δώσω το λόγο ε, και στην Ιρλανδική Προεδρία, στον Προεδρό της Σάμον Κόλλιν και μετά ε, στον Επίτροπο Τσούλος, Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα γεωργικά. Μετά από αυτά ε, θα ε, κάνουμε και μία πολιτική αξιολόγηση. Θα ζητήσω λοιπόν από τις πολιτικές ομάδες μέσω των συντονιστών τους να κάνουν μία πολιτική αξιολόγηση και ε, μετά το πέρας του γύρου των ε, συντονιστών θα δώσω το λόγο σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, όλους τους συναδέλφους που θα θελήσουν να πάρουν το λόγο. Ε, και βεβαίως κυρίως δίνοντας την προτεραιότητα σε αυτούς που θα έχουν διστάμενη άποψη από αυτή που θα έχει εκφράσει ο συντονιστής της ομάδος τους. Η τελική ψηφοφορία, επαναλαμβάνω, ότι θα ε, λάβει χώρα μετά την πλήρη γνώση των νομοθετικών κειμένων και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές. θα πρέπει να οργανώσουμε καλά τον χρόνο των αγοριτών και ε, το μάκρος των παρεμβάσεων, τη διάρκεια των παρεμβάσεων, ε, γιατί θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας μέχρι τις 5.30 σήμερα το απόγευμα, διότι αμέσως μετά ε, στις 5.30 δηλαδή, σε τούτη εδώ την ίδια αίθουσα, πάντα μαζί με τους εισηγητές, με τον εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας και με τον ε, κύριο Επίτροπο, θα δώσουμε συνέντευξη τύπου έτσι ώστε να παρουσιάσουμε την πολιτική αξιολόγηση. Με μεγάλη χαρά λοιπόν δίνω τώρα το λόγο στο Λουίς Κάπολο Σάντος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα δικά του θέματα πριν όμως του δώσω το λόγο να υπενθυμίσω σε όλους ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα επί των οποίων δεν έλαβε χώρα διαπραγμάτευση. Πρόκειται για θέματα τα οποία περιλαμβάνονται ε, στο ε, ε, διαπραγματευτικό box των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι θέματα επί των οποίων εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε γνώμη γιατί δεν έχουμε εντολή διαπραγματευτική επ' αυτών, άρα δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Αυτά τα σημεία ε, θα τα αφήσουμε στον διαπραγματικό γύρο των δημοσιονομικών προοπτικών, ευελπιστώντας ότι εκεί θα βρεθεί κάποια λύση. Εμείς ε, στην Επιτροπή Γεωργίας και στο Συμβούλιο Γεωργίας δεν μπορέσουμε να ανοίξουμε τα θέματα αυτά, γιατί δεν είχε εντολή το Συμβούλιο επί των σημείων αυτών. Ε, πρόκειται για συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει ήδη επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ε, εργάστηκαν για αυτό την δύσκολη διαπραγμάτευση ε, πάνω σε μια πρόταση της Επιτροπής η οποία τέθηκε σε αμφισβήτηση, η οποία ε, προκάλεσε πολλές διστάμενες απόψεις ε, και 8.000 περίπου τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους σκιώδης εισηγητές, τα 22 μέλη της Επραυτικής Ομάδας του Κοινοβουλίου, μαζί με την Προεδρία που σκληρά εργάστηκε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πολύ μας βοήθησε έτσι ώστε να επιτευχθούν συγκλήσεις από να ευχαριστήσω βεβαίως ε, και τον Γκέραλτ Κάλμπ από την γραμματεία που ξέρετε ότι θα μας αφήσει ε, τον ε, ε, Σεπτέμβρη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ολοκλήρωσε με τον τρόπο αυτό μία πάρα πολύ σημαντικό κύκλο εργασίας αλλά και τον Πάτρικ, την Ελένα, την, Ελένα, την Γετρούδη, όλους τους βουλευτές, συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ όλους για την εργασία σας και δίνω τον λόγο στον Λουίς Κάπολα Παρακαλώ. Ευχαριστώ Παόλο. Θα ήθελα Αρχικά, να χαιρετήσω τον Υπουργό Κόβενη. Σάιμον, καλώς Αγαπητέ Επίτροπε, Ντάτσιαν Τσόλος, αγαπητοί συνάδελφοι, Μόλις περατώσαμε μια, ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο στις εργασίες μας. Δεν περατώθηκε η εργασία μας και πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού. Ήταν μακρύτατη η διαδικασία και δυσχερέστατη ε, και πολλοί συνέβαλαν ε, σε αυτή την τελική επιτυχία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων που συνεργάστηκαν μαζί μου πάρα πολύ εντατικά και με αγαστό τρόπο. Σας ευχαριστώ ειλικρινέστατα. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα ήταν δυνατό να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα επίσης ε, να ε, ευχαριστήσω το τεχνικό προσωπικό, τη γραμματεία της Κόμα να ευχαριστήσω τη γραμματεία των πολιτικών ομάδων και την ε, Άννα Καμήλο, την γενική διευθύντριά μου, που είναι τόσο ικανή όσο και ολόκληρη γενική διεύθυνση. Ευχαριστώ την προσοχή σας στο ότι μελλοντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαθέτει ε, τα ίδια τεχνικά μέσα όπως το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έχουμε μεγάλες ανισότητες ως προς ε, το τεχνικό μας επιτελείο και ε, οι εργασίες μας ήταν ιδιαίτερα τεχνικές οπότε πρέπει να τονίσουμε παρκώς αυτό το σημείο. Ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων Όσοι γνωρίζουν τα αποτελέσματα θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την ε, διαπραγματευτική μας εντολή με ικανοποιητικό τρόπο. Ε, μας ανετέθη αυτή η διαπραγματευτική εντολή στο Στρασβούργο και τηρήσαμε την εντολή σχεδόν πλήρως. Κάναμε κάποιες παραχωρήσεις όπως εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και επικράτησε ένα πνεύμα συμβιβασμού και θέλω να το τονίσω αυτό για τα ουσιαστικά ουσιαστικά ζητήματα όμω για τι άμεσε ενισχύσει, ε, για το καθεστώ του ενεργού γεωργού, του μικρού γεωργού, του νέου γεωργού, για την εσωτερική σύγκληση, για την ε, ισότιμη κατανομή των ενισχύσεων, το greening, το πρασίνισμα. Πολύ δύσκολο ζήτημα. Ε, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ισορροπία, χάρη στο οποίο μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του οι γεωργοί, ενώ ταυτόχρονα τονίζουμε την πράσινη διάσταση που μας χαρακτηρίζει χαρακτηρίζει το οικολογικό τμήμα ενώ ήταν υποβαθμισμένο τώρα αυτό διαψεύδεται πλήρως από τα τελικά αποτελέσματα. Σε σχέση με τους πυλώνες θα σας πω ότι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο όπως παραδείγματο χάρη απαγόρευση των διπλών πληρωμών δεν θα υπάρξουν διπλές πληρωμές ε, πλέον στους γεωργούς και εισαγάγουμε με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη διαφάνεια και κυρίως μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον τομέα της γεωργίας ε, ενισχύοντας ε, τον πράσινο σε εισαγωγικά άξονα τη κοινή γεωργική ε, πολιτική, ε, σχεδόν ένα τρίτο του προϋπολογισμού διοχετεύεται προ αυτά τα μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, πράσινου χαρακτήρα. Δηλώνουμε όλοι ικανοποιημένοι όπως και οι σκιώδεις συζητητέ, Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια για τα όσα καταφέραμε. Ε, και ξαναλέω εδώ και τονίζω ότι αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη συνεργασία όλων των βουλευτών του Κοινοβουλίου και κυρίως των σκιωδών. Εν τέλει θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διάσταση που κρίνω αρνητική. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε σήμερα να κλείσουμε πλήρως αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, για να σας εξηγήσω γιατί δυστυχώς η Προεδρία έκρινε ότι δεν διαθέτει επαρκή διαπραγματευτική εντολή για να συζητήσει τα δημοσιονομικά ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε εντολή για μια συζήτηση όλη τη ύλη για την κοινή γεωργική πολιτική, καλύπτοντα όλε τι διαστάσει του ζητήματο. Δεν κατέστη δυνατό λοιπόν να αποφασίσουμε ουσιαστικά ζητήματα ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα και θα ε, αναπεμφθούν αυτά τα ζητήματα στην Επιτροπή μα. Ε, κατανοούμε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο Σάιμον. Είναι υπουργό Γεωργία, δεν είναι πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί τη χώρα του στο Υπουργικό Συμβούλιο και αντιμετωπίζει μεγάλε δυσκολίε δυσκολίες. Ε, θλίβομαι όμως που δεν μπορούμε να περατώσουμε τις διαπραγματεύσεις για όλα τα επιμέρους κεφάλαια της κοινή γεωργικής πολιτικής και αφήσαμε ε, πέρα αυτά τα ζητήματα δημοσιονομικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Ιδού. Ευχαριστούμε, Λουίς. Ο Μισελ Νταντάν τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Παύλο. Κοιτάξτε, μετά από πολλές ανταλλαγές ε, ε, ε, και συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων φτάσαμε σε μια συμφωνία όσον αφορά την κοινή οργάνωση των χωρών. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω προσωπικά την προεδρεύουσα χώρα, την Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν την αντίστοιχη και για την εργασία που κατέβαλαν αλλά και για το επικοδομητικό κλίμα μέσα στο οποίο εργαστήκαμε ο Λουίς ευχαρίστησε τη γενική του διευθύντρια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το δικό μου γενικό διευθυντή γιατί πραγματικά σε τέτοιου είδους θέματα ε, ε, στο Κοινοβούλιο βασιζόμαστε πάρα πολύ στους συνεργάτες μας γιατί δεν έχουμε και πολλούς άλλους ε, ανθρώπινους πόρους και γι' αυτό λοιπόν τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Κοινή οργάνωση αγοράς λοιπόν ήταν το θέμα που μας απασχολούσε. Ε, βασιζόμενοι σε δύο θέματα, ότι ε, θα έχουμε λιγότερους ε, πόρους, λιγότερα μέσα ε, έτσι, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε ε, να δοθούν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στις οργανώσεις παραγωγών ε, και στις οργανώσεις αγοράς έτσι ώστε να οργανωθούν καλύτερα. Μετά από την εργασία η οποία έλαβε χώρα, οι στόχοι που είχαν καθοριστεί στην εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούμε ότι οι όροι αυτής της εντολής έχουν γίνει σεβαστοί. Δεν ξεπεράσαμε γραμμές όπως άκουσα να λέγεται γίνεται δεξιά-αριστερά, αναφέρομαι κυρίως στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, αντιθέτως, εγγράψαμε ε, μία σειρά ε, αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων που θα έχουν πλέον οι οργανώσεις των παραγωγών και οι επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστότερη αντιμετώπιση του εισοδήματος των γεωργών σε μια αλυσίδα που γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια χάνει όλο και περισσότερο ε, την ε, ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα στις δύο άκρες αυτής της αλυσίδας. Ε, ήταν αρκετά ενωτική η γραμμή που ακολουθήσαμε δίνοντας τη μάχη αυτή και αυτό είναι ουσιώδου σημασία. Όσον αφορά τα μέσα υπάρχουν κάποια τεχνικά μέτρα, κάποια συμβολικού χαρακτήρα μέτρα και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε διατηρήσει μια η οποία όμως δεν βαραίνει ε, το, τα δημοσιονομικά. Αναφέρομαι κυρίως ε, στην ε, ζάχαρη. γιατί η ζάχαρη ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εξέβρεση συμφωνίας και αποφασίσαμε ότι μέχρι το 2017 θα εξακολουθεί το σύστημα των ποσοστώσεων ενώ στη βασική πράξη αναφερόμαστε στις συμβατικές υποχρεώσεις για την περίοδο μετά το 2017. Όσον αφορά τώρα τον αμπιλοεινικό τομέα προχωρήσαμε σε μία ε, καλή και ομαλή μετάβαση μέχρι το 2030. Αυτά που αποφασίσαμε ε, θα πρέπει τώρα ε, να τα εκμεταλλευτούν θετικά οι εμπλεκόμενοι φορείς. Δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο το οποίο θέτουμε στην διάθεση των γεωργών, των οργανώσεών τους, των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων και πρωταγωνιστών της γεωργικής αγοράς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της συμφωνίας τα οποία θα βελτιώσουν την προβλεψιμότητα της αγοράς, που θα επιτρέψουν ε, κοινέ δράσεις προς αποφυγή μελλοντικών κρίσεων. Εμείς, σαν πολιτικοί άνδρες και γυναίκες που, της πολιτικής, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την λειτουργία των μηχανισμών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πράξουν τούτο. Αλλά βεβαίως εμείς θα είμαστε ε, στην πορεία αρρωγή τους έτσι ώστε να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο είχε ο Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και από την δική μου πλευρά βεβαίως θα ήθελα ε, ως ήθιστε ε, αλλά και ουσιαστικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της ουσιαστικής συμφωνίας και που ήταν πάντα στη διάθεσή μας έστω ε, και προς ζημία της προσωπικής του ζωής ή άλλων προτεραιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την συμφωνία επί του θέματος αυτού. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσπαθήσαμε σκληρά και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν ε, συνεργάτες, ε, εισηγητέ, σκιώδεις κλπ. Στη διάρκεια λέω των διαπραγματεύσεων προσπαθήσαμε να μην ξεπεράσουμε καθόλου και να μην παρακάμψουμε την ε, εντολή που μας είχε δώσει η Ολομέλεια και να παραμείνουμε όσο γίνεται περισσότερο συνδεδεμένοι στο περιεχόμενο αυτής της εντολής. Βεβαίως αντισταθήκαμε στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Στο Λουξεμβούργο προημερών, δυόμιση ώρα τα ξημερώματα, ε, ε, βρισκόμαστε στην πιο διστάμενη δυνατή άποψη όσον αφορά ε, το φάκελο που μας ενδιαφέρει, αλλά έδειξαν καλή διάθεση Όλοι, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Κομισιόν έδειξε διάθεση να υποχωρήσει και τελικά ε, φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, ε, οι υπηρεσίες ε, και οι φορείς πληρωμής και αυτό ήταν ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Εμείς θέλαμε απλοποίηση και προσπαθήσαμε να την επιτύχουμε σε όλα τα περάσματα αυτές, αυτής της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής. Όσον αφορά τις υπηρεσίες τους φορείς πληρωμής, τελικά συμφωνήσαμε ότι οι, ελάχι, οι, ελάχιστες προσπάθειες ε, θα έπρεπε ε, να ε, οδηγήσουν σε μια τροποποίηση της παρούσας κατάστασης γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας των φορέων αυτών θα δημιουργούσε μεγάλα προσκόμματα στην καλή λειτουργία της κοινής γεωργικής Επίση, πολιτικής. Ε, επίσης ε, λέμε ότι θα πρέπει ένας οργανισμός, εθνικός οργανισμός πιστοποίησης να είναι σε θέση ε, να δώσει λύση σε όλες τις εσωτερικές διεργασίες των κρατών μελών. Εμείς αγωνιστήκαμε έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια των επιχειρηματικών συμβουλίων να μπορούν να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες ναι θα μπορούν μπορούσαν να είναι να αποφασίζονται κάθε φορά βάσει της βούλησης και των εργαζομένων ή των εμπλεκομένων φορέων αλλά λέμε ότι θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα. Ε, επίσης είχαμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά και την υλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, όσον αφορά τη λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σε πολλές περιπτώσεις είπαμε ότι μέσω κατεχώρηση πράξεων μπορεί το Κοινοβούλιο να ε, είναι ε, κύριος πρωταγωνιστής για την υλοποίηση της πολιτικής. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω το Συμβούλιο γιατί επί πολλών σημείων μας έδωσε την δυνατότητα να είμαστε πραγματικοί ε, πραγματικά παρόντες σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχία. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο η δημοσιονομική πειθαρχία γίνεται σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής. Θα έχουμε λιγότερα χρήματα, λιγότερους πόρους και επομένως ε, οι παρεμβάσεις αναθεώρησης προς τα κάτω, οι νέες υποχρεώσεις θα μας υποχρεώσουν να ε, έχουμε διαφορετική δημοσιονομική πειθαρχία. Επί του 25-2 επίσης ε, μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουμε πραγματικά στην εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας αντιταχθήκαμε στο Συμβούλιο, είμαστε αντιμέτωποι με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν σε πολλά θέματα, όπως ας πούμε την μείωση ή ε, την ε, διαγραφή των ε, ακύρωση των μηνιαίων πληρωμών. Εμείς σαν Κοινοβούλιο θέλαμε να δείξουμε, να, να, να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ε, γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε στις αναστολές πληρωμών. Εμείς αγωνιστήκαμε έτσι ώστε όπου είναι δυνατόν ε, και μέσα από πληροφορικές διαδικασίες να μπορέσουμε να έχουμε απλούστευση ε, ακόμα και μέσα από πολυετή αιτήματα. Προσπαθήσαμε να δείξουμε τι θέλει το Κοινοβούλιο όσον αφορά το Early Warning System, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ένα σύστημα δηλαδή το οποίο έγκαιρα θα δίνει την δυνατότητα να ταυτοποιηθούν απλά ε, ε λάθη, καθημερινά λάθη, ε, τα οποία μπορεί να διαπράττουν οι γεωργοί, έτσι ώστε να μην ξεκινάει για πολύ μικρά σφάλματα μια διαδικασία επί παραβάση. Επίσης, ε, σε πολλά άλλα ζητήματα έχουμε διαφορετική άποψη το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Κομισιόν, κυρίως όσον αφορά το θέμα του greening. Κοιτάξτε, εγώ έχω και πράσινη κάρτα, είμαι αναπληρωτής και έχω, είμαι και επισήμως πράσινος εδώ. Εν πάση περιπτώσει σας λέγω ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε ενδιάμεση λύση. Ευχαριστώ πάντω την Κομισιόν ε, γιατί μας έδωσε την δυνατότητα ε, στην αρχική φάση και της αρχικής εφαρμογής της πολιτικής αυτής ε, να ε, μας έδωσε λέω τη δυνατότητα να μην ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες επί παραβάση απέναντι στους γεωργούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Στους πρώτους δύο, ε, στα πρώτα δύο έτη εφαρμογής οι γεωργοί σε περίπτωση μη εφαρμογής του greening θα χάσουν μονάχα το, μέσο του, το, μέτρο του greening ενώ από το τρίτο έτος και πέρα θα έχουμε ε, την αύξηση σιγά σιγά του, του 25% μέχρι τη σταθεροποίηση του καθεστώτος. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα. Διαφάνεια, η υλοποίηση των ε, ε οδηγιών των ε, υδάτων και των αζωτούχων μια σειρά θεμάτων τα οποία οπωσδήποτε θα βοηθήσουν την ομαλή ροή της εφαρμογής της κοινή γεωργικής πολιτικής στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ όλους τους συζητητέ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ιρλανδική Προεδρία, στο Σάιμον Κόβενεν δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό. Για μία ακόμα φορά αισθάνομαι την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε ε, και ε, ε, την, μεγάλη δουλειά που έκανε γιατί πραγματικά ήταν τρομερό ισορροπιστή, Είχε 27 υπουργού από τη μία μεριά, 27 κράτη-μέλη από τη μία μεριά και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την άλλη. Thank you, Paolo. Ευχαριστώ Παύλο. και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής. Με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ τελευταίες μέρες της Ιρλανδικής Προεδρίας και είμαι στη θέση να κηρύξω την ολοκλήρωση μιας τελική συμφωνία για την κοινή γεωργική πολιτική και τη μεταρρύθμισή τη και, ένα πλαίσιο και την συζήτηση ενό πλαισίου σταθερού για τη γεωργική πολιτική και του γεωργού όλη την Ευρώπη, γιατί περί αυτού ακριβώ πρόκειται το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό για χρόνια. Έχουμε βέβαια περάσει από δύο οργανικές τριβές πρόκειται για μια νέα διαδικασία. Δεν έχει προηγηθεί άλλη συναπόφαση για την κοινή πολιτική στο παρελθόν. Δεν έχει προηγηθεί ε, διαπραγμάτευση με 27 σύντομα και 28 χώρες κατά την ολοκλήρωση διαδικασίας αναθεώρησης της ΚΑΠ στο παρελθόν. Και ως εκ τούτου είμαστε σε απάτητο έδαφος όλοι μας, αλλά έχουμε ευθύνη να φέρουμε αποτέλεσμα και το πιο σημαντικό πιστεύω για μένα, ο πιο σημαντικό τομέα ευρωπαϊκή οικονομία, η γεωργική πολιτική, τα τρόφιμα, η βιομηχανία τροφίμων εν γέννη. Και σε μια χρονική στιγμή όπου χρειαζόμαστε οι χώρες μας χρειάζονται νέα όθηση, βεβαιότητα, θέση εργασία και πάνω απ' όλα κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό που καταφέραμε τις τελευταίε τρει μέρε το ενέπνευσε η ανάγκη να αποδείξουμε ότι μπορούν σε εταιρική σχέση να συνεργαστούν τα θεσμικά μας όργανα και να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα για όλους τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε, γιατί περί αυτού τελικά πρόκειται. Να βρούμε έναν τρόπο, να φέρουμε αποτέλεσμα, να δώσουμε λύσεις σε δύσκολες περιστάσεις και μέσα στη, στη, στα βαθιά μεσάνυχτα και μέσα σε, από έντονες συζητήσεις, όπως επεσήμανε νωρίτερα και ο συνάδελφος, αλλά πάντως να βρούμε έναν τρόπο με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τα θεσμικά όργανα που εργάζονται με βάση αυτήν, να φέρουμε αποτέλεσμα για εκείνους που μας ψηφίζουν. Έτσι λοιπόν από τη δική μας την πλευρά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε μια πολιτική συμφωνία μετά από 43 διαπραγματεύσει τριμερού διαλόγου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάποιου μήνε μόνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πολύ σαφεί θέσει και πολύ σαφή εντολή, αγωνίστηκε σκληρά. Εξίσου όμω σαφή ήταν και δική, ήταν και δική μου εντολή εκ μέρου του Συμβουλίου. Αγωνίστηκα και εγώ να την ε, προαγάγω. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την αρχική τη θέση και διατήρησε όσο περισσότερο μπορούσε, όσο τη επέτρεπε η λογική να διατηρήσει από την αρχική τη θέση μέσα από τη διαδικασία αυτών των διαπραγματεύσεων. Και έτσι νομίζω ότι η επιτυχία, η πολιτική επιτυχία αυτής της ιστορίας είναι ότι αποδεικνύει πως μπορούν να φέρουν καλά αποτελέσματα για τους πολίτες στα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη, ακόμη και από περίπλοκες διαπραγματεύσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για τεράστια ποσά, 38% του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για το πρώτο έτος τουλάχιστον αντιστοιχεί στην ΚΑΠ. Για τη δική μου την ε, πατρίδα, είναι 7 χρόνια μιας δέσμης 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους Ιρλανδούς παραγωγούς, γεωργούς. Και βέβαια αυτό έχει και σημαντικές ε, δημοσιονομικές, ε, δημοσιονομικό αντίκτυπο. Πολύ μεγάλη πολιτική σημασία λοιπόν. Είχαμε ασφαλώς διασύνδεση και με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το δέχομαι. Εξού και έμειναν οι λεγόμενες αγγίλες ε, αναγκαστικά, το δέχομαι και αυτό. Δηλαδή όταν αποφασιστεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα κρυθούν κάποια ακόμα ζητήματα, αλλά Πάντω, για του γεωργού, για όσοι εκπροσωπούν εδώ την, γεωργική οικονομία και την ε, παραγωγή των τροφίμων εδώ, ε, έχουμε πλέον αποφασίσει και έχουμε επιλογέ για το πώ θα πληρώνουμε του γεωργού, πώ θα του ενισχύουμε, πώ θα δίνουμε την προτεραιότητα για τον νέο γεωργό, πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη μια νέα γενιά γεωργών ε, καλλιεργητών εκτροφέων που θα δίνουν τη δυνατότητα για παραγωγή τροφίμων πολύ πιο βιώσιμα, πολύ πιο οικονομικά, πιο, πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν και έχουμε επιτύχει μια ισορροπία για τα κύρια ζητήματα που απασχολούσαν τα θεσμικά όργανα. Όπως η διασύνδεση, που ήταν από τα πολύ δύσκολα προβλήματα του παρελθόντος και θεωρώ ότι έχουμε βρει μια συνετή συμβαστική λύση όσον αφορά την ενίσχυση στις αγορές όπου έχουμε διατηρήσει μια κίνηση προς ε, τις αγορές, τις ελεύθερες αγορές για τα τρόφιμα και την ε, γεωργία ε, τη γεωργική παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα με τη δυνατότητα επέμβαση όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Για το γάλα, το νίνο, τη ζάχαρη, ανάλογα με τις χώρες διαφορετικές προτεραιότητες, ανάλογα με τη χώρα διαφορετικές δομές, συστήματα προτεραιότητες και ε, συστήματα ενίσχυσης. νομίζω ότι βρήκαμε ισορροπίες που μπορούν να είναι ικανοποιητικές για τους πάντες. για την ευθυγράμμιση. Ε, κυρία Ρούντοστ και άλλοι που έχουν εμπλακεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα ότι ήταν πολύ δύσκολο το θέμα, δύσκολο και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να την επιλύσουμε, για να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστώ τον Λούις Κάπουλα Σάντος, τον Τζοβάνι Λαβία, τον Μισελ Ντοντάν, τον κύριο Ντεκάστρο, διότι για τη δουλειά που κάναμε όλοι μαζί τις τελευταίες εβδομάδες, ημέρες, μήνες και όλους τους άλλους. Όλοι όσοι έλαβαν μέρος ως ε, εισηγητές και εισηγητές, ε, από, άλλες πολιτικές, από όλες πολιτικές ομάδες, όλοι όσοι συνέβαλαν στην διαδικασία αυτή από πλευρά του Κοινοβουλίου και ήταν καθοριστική η συμμετοχή σας. Και πρέπει να πω ότι ως πρώην Ευρωβουλευτής ε, πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο αποδεδειγμένα έχει εξασφαλίσει την το δικό του σημάδι, έχει βάλει το δικό του σημάδι σε αυτή τη μεταρρύθμιση, το σημάδι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λέω αυτό εκπροσωπώντας και το Συμβούλιο που καλούμε να εκπροσωπήσω, που οφείλω να εκπροσωπήσω ως ε, εκπρόσωπος Προεδρίας. Για το greening, το πρασίνισμα, το οποίο είναι ένα θέμα σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ίσως και το πιο σημαντικό δείγμα αλλαγής πολιτικής μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση. Δύσκολο θέμα, δυσεπίλητο. Θελήσαμε να δώσουμε απλές λύσεις, αλλά ταυτόχρονα με σαφέ πλεονέκτημα για το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος με την εισαγωγή των μέτρων του πρασινίσματος. Τώρα έχουμε ορόσημο εγγύηση για τον πρώτο πυλώνα, όπου όλοι οι γεωργοί θα πρέπει να ξεπερνούν το ορόσημο αυτό για να εξασφαλίσουν τι πληρωμές του πρασινίματο τώρα και στο μέλλον να αποφεύγουν τι. Στο δεύτερο πυλώνα επιπλέον τα κράτη θα κάνουν και άλλα πράγματα όταν θα θέλουν να δώσουν προτεραιότητε ανάλογα με τι κλιματικέ του συνθήκε, τα, τα είδη των καλλιεργειών, τη γεωφυσική του κατάσταση και το Και έτσι μπορούμε πιστεύω πια όλοι από κοινού να υπερασπιστούμε μια ισορροπημένη και προοδευτική μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής που θα προστατεύει το περιβάλλον καθώς έχουμε καθήκον να το πράξουμε αλλά και θα επιτρέπει επίσης και την ανάπτυξη και την επέκταση στον ε, τομέα αυτών για το μέλλον σε μια περίοδο όπου ολόκληρος ο κόσμος και η Ευρώπη ιδιαίτερα χρειάζεται να μπορεί να παράγει τρόφιμα κατά τρόπον αιφόρο. Έτσι και στην κατανομή των ποσών εσωτερικά ήταν πολύ σημαντικό για μένα να εξασφαλίζω ότι θα μπορούν οι χώρες να έχουν επιλογή στην αναδιανομή των ποσών έτσι ώστε η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη στους τομείς τους ανάλογα με την περίπτωση να, εξασφαλίζεται, να εξασφαλίζεται και ταυτόχρονα βέβαια να είναι πιο δίκαιη η κατανομή των ενισχύσεων σε αυτούς που τη χρειάζονται. Αισθάνομαι λοιπόν και ανακούφιση και ικανοποίηση που μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αυτή. Μια δουλειά που ξεκινήσαμε τον προηγούμενο Γενάρη και πιστεύω ότι ε, απαντούμε στις προσδοκίες των γεωργών, των παραγωγών, της βιομηχανίας τροφίμων με τις προσπάθειές μας της τελευταίας εβδομάδας. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον Επίτροπο κύριο Τσόλος, ο οποίος ήταν ο κινητήριος, ε, ήταν ο κινητήρας της διαδικασίας αυτής. Ε, πολλές φορές χρειάστηκε σαν το διαιτητή να σφυρίζει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αλλά και που ταυτόχρονα έχει ένα σεφάστατο όριμα, για το τι θέλει να επιτύχει και τη μελλοντική μεταρρύθμιση, για το μέλλον της μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ και έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτήν. Και μια και, από ό,τι φαίνεται, μια φορά μπορώ να τα πω όπως θέλω, θέλω να ευχαριστήσω τη δική μου ομάδα, να ευχαριστήσω τη δική μου ομάδα που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην Ιρλανδική Προεδρία και ο Λουίς το επεσήμανε, ότι οι πόροι που έχει στη θέσή του ένας ευρωβουλευτής μερικές φορές περιπλέκουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τη συναπόφαση. Και αληθεύει αυτό όντω, γιατί και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ ευρωβουλευτής και καθόμουν στα έδρανα όπως εσείς. Είναι μεγάλες ε, οι δυνατότητες που μπορεί, από τις οποίες μπορεί να αντλήσει πόρους ο Ευρωβουλευτής, ενώ εγώ από το Υπουργείο Γεωργίας της Ιρλανδίας ως προεδρεύων είχα πολύ περιορισμένε δυνατότητε και γι' αυτό και φίλω θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτε μου που κατέστησαν δυνατή αυτή την επιτυχία και βέβαια και στη γραμματεία του Συμβουλίου που συνέβαλε τα μάλα στι προσπάθειε αυτέ και στην επιτυχία. Και πάλι λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου εδώ στο Κοινοβούλιο για την υποστήριξη, για τη συνεργασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τώρα όλοι να βγούμε και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε την αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, η προοδευτική μεταρρύθμιση τη κοινή πολιτική που θα χαράξει το σημάδι τη πάνω στην Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή για την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Σάιμον. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο υπεύθυνο για θέματα γεωργία, τον κύριο Τσιόλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από τρία χρόνια περίπου, Θα θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει μια, ένα δημόσιο διάλογο για τη μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής. Τρία χρόνια μετά λοιπόν, να είμαστε που ξανά είμαστε εδώ μπροστά σα, οι ενώπιον ημών των ε, νομίμων και ερετών εκπροσώπων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμαστε λοιπόν να σας δώσουμε τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά μιας μεταρρύθμισης, η οποία πια φτάνει στην ολοκλήρωσή της, ύστερα από ένα δημόσιο διάλογο, ύστερα από μια μεταρρύθμιση ανοιχτή στην κοινωνία και που στόχο είχε να προσφέρει στον Ευρωπαίο Γεωργό τα μέσα να επιτελέσει το έργο του έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό το άνοιγμα της γεωργικής πολιτικής προς την κοινωνία της Ευρώπης που θελήσαμε εμείς να διαφυλάξουμε, να εξασφαλίσουμε, ε, συνεπάγεται βέβαια πολύ πιο περίπλοκη δουλειά για τον γεωργό, τον παραγωγό, συνεπάγεται πολύ περισσότερε προσδοκίες που επομίζεται και νομίζω ότι αυτή η περίοδος της μεταρρύθμισης και, και τα μέσα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τον γεωργό και τον παραγωγό για να είναι πιο ε, παραγωγικός για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες της κοινωνίας και να φέρουν αυτή τη στιγμή την, ε, ε, να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή της ανταλλαγής και της επικοινωνίας της κοινωνίας με τον Γεωργό και τον Παραγωγό. Για το Κοινοβούλιο, νομίζω, ως συνομοθέτη, ήταν ο πιο φυσιολογικός ρόλος να εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Μια κοινή γεωργική πολιτική, λοιπόν, μεταρρυθμιζόμενη, μεταρρυθμισμένη, η οποία χαρακτηρίζεται, πιστεύω, από ένα κοινό πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα και από την πραγματικότητα που διαβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, 27 και σύντομα 28 κράτη-μέλη συγκεκριμένα, που με μια κοινή γεωρική πολιτική ηλικίας 50 ετών και που υποχρεούνται να δώσουν, υποχρεούνται να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις για τη διαχείριση των 400 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ του Ευρωπαίου Φορολογουμένου για τα 7 προσεχή έτη. Και πολύ σωστά ε, έρχεται μερικές φορές ο πολίτη να ρωτήσει τι, σε τι χρησιμεύει αυτός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Να λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα σε τι πηγαίνει, σε τι χρησιμεύει το 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, και πρέπει να βρούμε όχι μόνο τρόπο να διαχειριστούμε χρηστά αυτά τα ποσά, αλλά και να τα κάνουμε ορατά και κατανοητά το πώς διαχειριζόμαστε και πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά για τον Ευρωπαίο πολίτη σήμερα. Η κοινή γεωργική πολιτική λοιπόν μεταρρυθμισμένη και καταγράφοντας και καταγράφει το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο το εδαφικό, τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με όλα τα στοιχεία της ευελιξίας που ενσωματώθηκαν σε αυτήν τη νέα γεωργική πολιτική, αλλά και τις δομές της παραγωγής και της, ε, των προσανατολισμών της παραγωγής, τις ιδιαιτερότητες τις τοπικές, ε, οι οποίες ε, ενσωματώνονται στις διάφορες επιλογές που έχουμε καταθέσει στις προτάσεις. Κύριε Επίτροπε, μου λένε πολύ συχνά, εσείς Κοινοβούλιο, εσείς Συμβούλιο, ε, μου λέτε η μεταρρύθμισή σας μα ζητάει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Όχι, θα σα εξηγήσω. Ακριβώς αυτό είναι νομίζω το κύριο στοιχείο αυτής της μεταρρύθμισης, το ότι εμπλέκεται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και έτσι χάρη σε αυτά δίδονται κατευθύνσει μια κατεύθυνση που από την αρχή επελέγει ευρωπαϊκή ε, κατεύθυνση με κοινά μέσα, με κοινού στόχου που με αλλαγές κάποιων κανόνων στην πορεία επιτρέπουν την επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών στην κάθε χώρα, στην κάθε περιοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολύ πιο καλά εστιασμένη γεωργική πολιτική τώρα, με συγκεκριμένες κατηγορίες γεωργών που χρειάζονται την ενίσχυση, είναι πολύ πιο δίκαιη η νέα πολιτική γιατί έχουμε και πιο σαφή, πιο ισότιμη και πιο διαφανή κατανομή των ποσών που χορηγούνται στους ε, παραγωγούς. Είναι πιο πράσινη η γεωργική πολιτική και ταυτόχρονα μπορεί να προχωρήσει σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα για τον γεωργό και τον παραγωγό. Και προχωρώ πολύ γρήγορα στα όσα έχουμε επιτύχει μετά την ε, υποβολή της νομοθετικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περίπου 50 τριμερών διαλόγων, περίπου 50 τριμερείς συνεδριάσεις Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τελευταίο μήνα. Για τις άμεσες ενισχύσεις λοιπόν έχουμε σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών, εξωτερική δηλαδή, και εσωτερική σύγκληση, η οποία εν τέλει επιτρέπει την ευελιξία και τις επιλογές για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, ώστε ακριβώς αυτή η σύγκληση, αυτή η κατανομή, η πιο ισότιμη κατανομή των ενισχύσεων για το γεωργό να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις διαφορετικέ ιδιαιτερότητες αλλά και τις ιδιαιτερότητες ανάλογα με τον τύπο της γεωργικής παραγωγής ή τον τύπο της γεωργικής εκμετάλλευσης διότι έχουμε ένα ελάχιστο κατόφλι σύγκληση που καλύπτει τι χαμηλότερε ενισχύσει, των οποίων τα ποσά θα αυξηθούν στα προσεχή έτη, αλλά και που ταυτόχρονα ορίζει ε, περιορισμό των απολειών για εκείνους που είχαν περισσότερα τώρα, έτσι ώστε η μείωση των ενισχύσεων για αυτή την κατηγορία να μην θέσει σε κίνδυνο την οικονομική τους επιβίωση η βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα όμω υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να περιφερειοποιήσουν αυτέ τι ενισχύσει, λαμβάνοντα υπόψη ομοιογενή περιοχή γεωργικού χαρακτήρα, οικονομικού ή διοικητικού. Μια διαδικασία λοιπόν σύγκληση των άμεσων ανισχύσεων ε, που θα είναι πιο προσαρμοσμένε στι πραγματικότητε τη κάθε περιοχή, του κάθε κράτου και ήταν αυτό μεγάλη προσδοκία και απέτηση των κρατών στο θέμα αυτό, το γνωρίζω. Επίση λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητε των νέων κρατών μελών τα οποία για μια μεταβατική περίοδο μπορούν να διατηρήσουν τα ειδικά συστήματα ενισχύσεων κατά, ε, αναέκταση, όπως είχε προταθεί το σύστημα κατά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα τις ενισχύσει αυτές να τις συμπληρώνουν από τον εθνικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχουν φτάσει τον ευρωπαϊκό μεσόρο των ενισχύσεων, έστω και αν αυτές οι πληρωμές θα αυξηθούν τα προσεχή έτη και έτσι θα πλησιάσουν το μεσόρο τη της Έχουμε ταυτόχρονα έναν ορισμό του ενεργού γεωργού με έναν αρνητικό κατάλογο, κατάλογο αποκλεισμού δηλαδή για, ορισμένους, για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων που ξεκάθαρα δεν είναι ενεργοί γεωργοί. Έναν ορισμό λοιπόν ανεγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ταυτόχρονα δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προσθέσουν, να συμπληρώσουν στον κατάλογο αυτό και άλλες κατηγορίες έτσι ώστε να λάβουν υπόψη τους ιδιαίτερες ε, συνθήκες ε, που χαρακτηρίζουν για τα κράτη αυτά τον ενεργό γεωργό. Και έχουμε επίσης και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό ένα μέσο το οποίο ιδιαίτερα απευθύνεται στον νέο γεωργό ε, στον πρώτο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής μάλιστα, εκεί όπου μιλούμε για άμεσες ενισχύσεις. Και έτσι έχουμε όχι μόνο το μέσον της Ανάπτυξη της υπαίθρου που απευθύνεται στο νέο με την ενίσχυση για την εγκατάσταση κτλ. αλλά και που προτείνει για τα πέντε πρώτα χρόνια από την εγκατάσταση οικονομική ενίσχυση για τον νέο ε, γεωργό. Και εδώ ευχαριστώ ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο απεδέχθη αμέσως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια οφείλω ευχαριστίες και προς τη φρόνηση του Συμβουλίου των Υπουργών που εν τέλει εδέχθη αυτήν την πρόταση. Ξέρω ότι ο Σάιμον Κόβενι εκπροσωπώντας βέβαια πάντα όπως όφιλε και πολύ καλά μάλιστα την, ε, τις θέσεις του Συμβουλίου, ο ίδιος προσωπικά ήταν επεπισμένος για την ανάγκη να δοθούν αυτές οι ενισχύσεις προς τους νέους γεωργούς και χάρη και σε αυτόν μπορέσαμε να επιτύχουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ενίσχυσης των νέων γεωργών ιδιαίτερα. Για καταστάσεις ιδιαίτερες διαφυλάξαμε τις συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις για να διατηρήσουμε για ορισμένες περιοχές ε, και κατηγορίες και τομείς την υποστήριξη εκεί όπου έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ε, σταθερότητα, για την εδαφική ισορροπία σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Και έχουμε ένα 30% των άμεσων ενισχύσεων που εκπροσωπεί μάλιστα το μεγαλύτερο τμήμα της κοινή πολιτικής σε, που μετακυλούνται σε πρακτικές γεωργικές όχι μόνο βιώσιμες αλλά ταυτόχρονα εντασσόμενες μέσα σε ένα στόχο ανάπτυξης και παραγωγής γεωργικής αηφόρου από πλευράς του γεωργού και βέβαια με βάση τις συζητήσει που κάναμε τα τελευταία χρόνια τον τελευταίο 1,5 χρόνο καλύτερα και τους τελευταίους μήνες πιο συγκεκριμένα μπορέσαμε να βρούμε λύσεις ε, για το πρασίνισμα που βοηθούν αυτούς που ήδη κάνουν, έχουν βρει λύσεις για το πρασίνισμα, που δεν θέτουν σε δυσμενέστερη θέση εκείνους που έχουν βρει λύσεις για το πρασίνισμα, που μεριμνούν για την ανάπτυξη μιας γεωργικής παραγωγής με ποιότητα και ε, βιωσιμότητα και αηφορία και που ταυτόχρονα βοηθούν στην ανάπτυξη αηφόρων γεωργικών πρακτικών. Επίσης, καταβάλαμε ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι μικροί γεωργοί και να τους δώσουμε την δυνατότητα να φτάσουν στην αγορά, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ε, και των ε, πολιτών καταναλωτών και των πολιτών ε, φορολογουμένων δημιουργούμε ένα απλουστευμένο σχήμα στις χώρες μέλη στον πρώτο πυλώνα που στηρίζει μέσα από σειρά ε, μέτρων της ανάπτυξης ε, της υπαίθρου που μεταξύ άλλων στηρίζουν και την τοπική αυτή παραγωγή. Ε, όσον αφορά τον ε, κανονισμό διαχείρισης ε, της και οργάνωσης της αγοράς. Εμείς μειώνουμε τον ρόλο της γραφειοκρατικής παρέμβασης του δημόσιου τομέα που συχνά δυσκολεύει τη διαχείριση της αγοράς. Αυξάνουμε την εμπλοκή των ε, επαγγελματικών οργανώσεων των ε, παραγωγών και ε, με την στήριξη του Κοινοβουλίου το αναγνωρίζω και κάποιων τροπολογιών του Κοινοβουλίου αλλά και με τη στήριξη του Συμβουλίου μπορέσαμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς διαχείριση κρίσεων που συχνά καταστρέφουν τους γεωργούς ε, παρά δηλαδή μια καλή διαχείριση των οικονομικών τους και της δραστηριότητάς τους ε, μπορεί να πέσουν έξω μέσα από τέτοιου είδους κρίσεις ε, και επομένως δίνουμε περισσότερα εργαλεία στους ίδιους τους γεωργούς να διαχειριστούν τις εν λόγω αλλά και στους διαχειριστικούς φορείς δίνουμε την δυνατότητα να βοηθήσουν τους γεωργούς σε στιγμές ακριβώς επίγουσας ανάγκης ολοκληρώσαμε ε, την ε, δέσμη γάλακτος που είχε αποφασιστεί πριν από λίγο καιρό ε, και καταφέραμε να φτάσουμε και σε μία τροποποίηση, μία μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης, λαμβάνοντας υπόψη το τέλος των ποσοστώσεων της ζάχαρης σε μια λογική χρονική περίοδο. Και τέλος προτείναμε και ένα νέο εργαλείο για τη διαχείριση του εμπελιονικού τομέα έτσι ώστε η πλαισίωση των ε, ε, καλλιεργημένων επιφανειών του εμπελονινικού τομέα ε, να δώσει την δυνατότητα προστασίας της παραγωγής αλλά και προστασίας των εδαφών. Μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία και για τις περιφέρειες και για τα κράτη-μέλη αλλά και συγκεκριμένες ε, προτεραιότητες ε, που αφορούν την ε, δυνατότητα παραγωγής, την ποιότητα παραγωγής, την διαφοροποίηση της παραγωγής που ενισχύει επίσης και ενθαρρύνει τους γεωργούς να οργανωθούν και να συμμετάσχουν λοιπόν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Και τέλος ε, με τον οριζόντιο κανονισμό ε, και χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των τροπολογιών του Καταφέραμε, λέω, να φτάσουμε σε μια γεωργική πολιτική ε, της οποίας η διαχείριση θα είναι καλύτερη γιατί ε, δεν θέλουμε απλώς να ε, προσανατολίσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων σε σωστή κατεύθυνση αλλά έχουμε ενισχυμένα εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων αυτών και μια γενικότερη κοινή γεωργική πολιτική που θα είναι και πιο απλή για την διοίκηση και για τους γεωργούς αλλά και πιο διαφανής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ολοκληρώνεται μια διαδικασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο ε, Παολό Κάστρο, ο οποίος ε, ορθότατα διαχειρίστηκε αυτήν την εμπλοκή, την πρώτη εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην διαδικασία στην απόφαση. τον Λουίς Μανουέλ, ε, ο οποίος ήταν εισηγητής για δύο από τους σημαντικότερους κανονισμούς αυτής της μεταρρύθμισης και που πέρασε ολόκληρες μέρες και νύχτες καθόλου εύκολες. Ε, ξέρω ότι τον τελευταίο καιρό ε, προσπαθούσε να εκπροσωπήσει όσο γίνεται καλύτερα τις προσδοκίες των συναδέλφων του ε, μελών του Ευρωπαϊκού Βουλίου. Ευχαριστώ πολύ τον Μισελ κυρίως για την δυναμική του και επικοδομητική του εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για έναν ε, κανονισμό ο οποίος ήταν πολύ δύσκολος ε, και ενέπλεκε διαφορετικές προσδοκίες ε, της κάθε πλευράς. Να ευχαριστήσω και τον Τζοβάνι γιατί αντιμετώπισε ένα δύσπεπτο οριζόντιο κανονισμό που όμως τελικά πολλά καλά θα φέρει στην κοινή γεωργική πολιτική. Τέλος, να ευχαριστήσω τον τον Σάιμον γιατί υπό Ιρλανδική Προεδρία και κάτω από την δική του καθοδήγηση καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την μεταρρύθμιση. Ο Σάιμον είναι ένας νέος πολιτικός άνδρας από αυτούς που θα ήθελαν να υπάρχουν περισσότεροι στον πολιτικό βίο. Από κάθε άποψη ήταν ευχαρίστηση να δουλέψω μαζί του, αλλά κυρίως τύχη, πολύ καλή τύχη για την κοινή γεωργική πολιτική ε, που βρισκόταν ο Σάιμον ε, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης από Ιρλανδικής πλευράς λοιπόν είχαμε το Σάιμον σε αυτή την πολύ αποφασιστική στιγμή. Θα ήθελα και ενώπιόν σας να ευχαριστήσω τους, συναδέλ συνεργάτες μου της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη που ήταν πάντα ε, στο πλευρό μου. Ξεκινήσαμε το 2010 και ολοκληρώσαμε τώρα, αλλά βεβαίως ε, η εργασία μας δεν τελειώνει εδώ, γιατί αν τώρα μας δώσετε εντολή θα ξεκινήσουμε και την ε, προσπάθεια υλοποίησης και την προετοιμασία της υλοποίησης αυτής της μεταρρύθμισης. Ε, γιατί θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας ε, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Και η κοινή και η κοινή πολιτική που θα προκύψει θα ανταποκρίνεται και αυτή στις προσδοκίες σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Ευχαριστώ πολύ και τον Ντάτσεν Τσόλος. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων περιμένω βεβαίως από πλευράς τους πολιτικές αξιολογήσεις. Όπως είπα και προηγουμένως δεν θα ζητήσουμε εν τέλει ψηφοφορία αλλά πολιτική αξιολόγηση. Ε, θα περιμένουμε την έγκριση των ε, δημοσιονομικών προοπτικών για να μιλήσουμε για τα οικονομικά. Ε, τώρα θα ξεκινήσουμε από τον Άλμπερντ Ντες βεβαίως μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον Λουίς Κάπολα Σάντος εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και σιγά σιγά θα δώσω το λόγο σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Άλμπερτ δεν έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ Παόλο, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι εισηγητές, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα, ύστερα από χρόνια διαπραγματεύσεων, από πολυάριθμες ακροάσεις, συζητήσεις, 8.000 τροπολογίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο μας για τη μεταρρύθμιση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλω ευχαριστίες προς όλους τους εμπλεκομένους, εισηγητές και όδη εισηγητές, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, από σε σένα Σάιμον, στον κύριο Επίτροπο, όλο το προσωπικό που συνεργάστηκε σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Το αποτέλεσμα προσφέρει βεβαιότητα και δυνατότητα προγραμματισμού για όλους τους γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οικογένειές τους μέχρι το 2020 και ταυτόχρονα προσφέρει ένα αποτέλεσμα την, αηφόρο, την πιο αηφόρο γεωργία της, του κόσμου να την κάνουμε ακόμη πιο αηφόρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρόκειται για ένα αποτέλεσμα το οποίο σημαίνει ότι ταυτόχρονα μπορούμε να ε, προσφέρουμε και υψηλής ποιότητας ε, τρόφιμα για τα εκατομμύρια των πολιτών, εκατοντάδες εκατομμύρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμβασμοί βέβαια πάντα είναι συμβασμοί, ε, σημαίνουν δηλαδή συγκερασμό διαφορετικών θέσεων. Ο συγκερασμός των θέσεων της, ε, του γεωργικού κόσμου των 27 κρατών μελών ε, ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν κοινέ θέσει. Συμβασμό βέβαια σημαίνει ότι κανεί ποτέ δεν έχει ασφαλίσει το 100% των απαιτήσεων ή προσδοκιών του και ταυτόχρονα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπό την Ιρλανδική Προεδρία με του δικού μα εισηγητέ, με τον ε, αξιότιμο πρόεδρο τη Επιτροπή μα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αποδεκτό για όλους μας πιστεύω. Έκανα μόλις μία συνεδρία με την ομάδα ε, γεωργικών θεμάτων της, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμπεραίνουμε όλοι οι συνάδελφοι μαζί ότι εν γέννη μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τις ε, συμβαστικές αυτές προτάσεις. Ξέρετε, ε, λέμε στη, στο χωριό μου, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, όταν περάσει μια πολύ δύσκολη μπόρα, ε, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Έτσι λοιπόν και τώρα, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την πρόταση, από αυτή τη συμβαστική πρόταση. Και κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο στην ευρωπαϊκή ιστορία να έχει γνωρίσει μια νομοθετική διαδικασία 8.000 τροπολογίε. Ένα θετικό νομίζω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ότι όλοι οι συνάδελφοι πλάκησαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία της μεταρρύθμισης και αξιοποίησαν τις ε, διατάξεις και τις προβλέψεις ε, της συνθήκης Λισαβόνας γιατί τις πήραν πολύ σοβαρά υπόψη. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να φροντίσουμε η, ε, τα συμπεφωνημένα να τηρηθούν, να υλοποιηθούν και να περάσουν πλέον στην διαδικασία της υλοποίησης και βέβαια της αποδοχής από αυτούς τους οποίους αποσκοπεί, στους οποίους στρέφεται και απευθύνεται αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό παρακαλώ στο δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία κατά την εκτέλεση. Η γεωργία στην Ευρώπη είναι ο τομέας του μέλλοντος. Η γεωργία είναι ένας τομέας θετικός και γι' αυτό θα ήθελα να πω ήδη σε αυτό το σημείο Γνωρίζοντα ότι μας παρακολουθεί η κοινή γνώμη ότι αν έχουμε το 40% αυτό του ευρωπαϊκού προπολογισμού αφιερώσει στην, στην ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να ξέρουμε γιατί έχουμε τόσο αυτό το 40% διότι κανένα άλλο τομέα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είχε μπορέσει να ε, δώσει τέτοια αποτελέσματα όσο αυτός της γεωργίας. Ότι αν, είχε ρυθμιστεί, αν είχαν ρυθμιστεί όλοι οι άλλοι τομείς της ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτικής όπως ο γεωργικός τομέας, τότε δεν θα είχε μείνει ούτε 1% για τη γεωργία από το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε, πάνω απ' όλα πρέπει να δώσουμε προοπτικές για τον πρώτο αλλά και από τον δεύτερο πυλώνα για την νεολαία μας, για τη νέα γενναία των γεωργών και Βεβαίω θα ακούσω και του συναδέλφου. Πάντω θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρόκειται να υποστηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση. Έχουμε τουλάχιστον την πολιτική υποστήριξη εκφράσει για τη δικασία αυτή τη μεταρρύθμισης και θα την παρακολουθήσουμε επικοδομητικά. Εμεί στο Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα και χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα να παρακολουθήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη τη υπόθεση αυτή και θα ήθελα εδώ να κάνω μια προσωπική ε, παρατήρηση. Εγώ ξεκίνησα την, ε, τις σπουδές μου στη γεωπονική την ώρα που ξεκινούσε και η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρώπης, δηλαδή 50 χρόνια πριν. Και δεν ξέρω αν εγώ παρακολουθώ τη γεωρική πολιτική ή αν εκείνη με ακολουθεί κατά πόδαν. Πάντω έχω προχωρήσει μαζί με τη γεωρική πολιτική τη Ευρώπη και μπορεί πιστεύω αυτή η γεωρική πολιτική να συμβάλλει όπω και στο παρελθόν σε ένα σαφέ, ε, στο να καταστεί ένα σαφή παράγον ενοποίηση τη ευρωπαϊκή διαδικασία. Χωρί αυτή την κοινή γεωρική πολιτική ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα έχει επιτευχθεί, τουλάχιστον στου όρου στου οποίου έχει επιτευχθεί αυτή η ενότητα, αυτή η ενοποίηση τη Ευρώπη, αυτή η ολοκλήρωση δηλαδή και αυτήν πρέπει να τη διαφυλάξουμε πιστεύω πιστεύω, ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συνέπραξαν στην υπόθεση αυτή και πιστεύω ότι μπορούν όλοι οι γεωργοί της Ευρώπης να είναι ικανοποιημένοι με, αυτές τα, με αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Ο Λουί Κάπουλα Σάντο, όχι σαν εισηγητή, αλλά σαν συντονιστή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πάολο. Από τότε που έγινε η σύσκεψη στο Λουξεμβούργο, η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μπόρεσε στην Ολομέλεια τη ομάδα να κάνει μια ευρύτατη συζήτηση και κάναμε και δύο συσκέψεις τη ομάδα εργασίας για την Γεωργία. Και από τι αντιδράσει των συναδέλφων σε όλε αυτές τις συσκέψει. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια εξαιρετικά ευρεία συνένεση για τα ε, πορίσματα των διαπραγματεύσεων και επισήμως ε, ε, απεφάνθη η ομάδα. Σε δύο μέρες έγιναν τρεις συσκέψεις και είναι ευμενείς οι αντιδράσεις των σοσιαλιστών και δημοκράτων. Ο συνάδελφος Λάιον από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Θυμηθείτε το 2010 όταν άρχισε η Επιτροπή να συζητάει τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής, φαίνεται να έχει περάσει μια ζωή από τότε. Σε αυτή την ε, έκθεση που συνέταξα εγώ προς μεγάλη μου τιμή και εγκρίναμε τότε, ποιο ήταν το ζητούμενο, ότι εν ώψη των μεγάλων προκλήσεων ε, του αυξανόμενου πληθυσμού και της αυξανόμενης ζήτησης για τροφή, πώς θα μεριμνήσουμε τόσο ώστε να γίνει βιώσιμη κοινή γεωργική πολιτική για να παράξουμε περισσότερο φαγητό χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Σήμερα το ζητούμενο ε, είναι να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η βιωσιμότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι στον πυρήνα της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, και θα αποτελέσει κίνητρο και θα ανταμείψει μια παραγωγικότερη γεωργία που παράγει περισσότερα και χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους στο μέλλον. Πιστεύω μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ε, μας κατέκριναν ότι ασχολούμαστε υπερβολικά με τη βιοπικιλότητα και την ε, αποτελεσματικότητα των λοιπασμάτων, ε, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων όλα αυτά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση την επιθυμητή να ταΐσουμε όλους αυτούς που θα πεινάσουν στο μέλλον χρησιμοποιώντας ε, ε, λιγότερους πόρους. Έχουμε τους ε, νέους γεωργούς, τους ενεργούς γεωργούς, τα περιβαλλοντικά μέτρα είναι μια σειρά πάρα πολύ θετικών μέτρων που θα κατοχυρώσουν την παροχή δημοσίων επισητιστικών αγαθών στο μέλλον και άρα πιστεύω ότι στον πυλώνα 1, η μεταρρυθμιστική πολιτική εξυπηρέτησε τον επιδιωκόμενο στόχο τι τελευταίε 200 ώρε και ακούω αποκλίνουσε απόψει. Πώ ήταν αυτή η τριμερή διάλλαγη. Ο Σάιμον είπε 42, ο Επίτροπο είπε σχεδόν 50. Ε, ε, ωραία, α κάνουμε ένα συμβασμό. 46 α πούμε ότι ήταν η τριμερή. ε, τις ε, περασμένες 8 εβδομάδες ε, δείξαμε ότι πραγματικά λειτουργεί η διαδικασία συναπόφασης ε, γιατί έδωσε ένα αυτό αποτέλεσμα και η γεωργοί και η αγροβιομηχανία αυτό περίμεναν. Μας ε, ρωτούσαν πότε τελικά θα καταλήξετε σε ένα πακέτο που θα μας πει τι μέλη γενέστε και ποια συστήματα ενισχύσεων, με ποια συστήματα ενισχύσεων θα πρέπει εμείς να συμμορφωθούμε. Τους δώσαμε όμως τη γενική γραμμή και αυτή είναι η γραμμή της βιώσιμης ε, γεωργίας για τη μελλοντική γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω γιατί όλοι ενέργησαν με ε, ιδιαίτερα επαγγελματική στάση. Ε, μιλώ και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο και για την, τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Προεδρίας, τον Υπουργό Κόβενη. Οι εισηγητές τώρα και οι σκιώδεις Σε κάθε φορά που συσκεπτόμασταν το Συμβούλιο είχε 20 αξιολογικές από πίσω που του έδιναν συμβουλές. Εμείς ε, είχαμε κάποιους ε, συμβούλους ε, λιγοστούς. Είναι μεγάλη ανισότητα και για να καταστήσουμε πιο επαγγελματική τη μεθοδολογία εργασίας μας θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογές για να μπορούμε να ακολουθήσουμε και το ρυθμό που μα ζητάτε. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμίσουμε τέλο. Η μοναδική επίκριση που έχω να απευθύνω είναι για τα διαπραγματευτικά κουτιά του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είχαμε το αποθεματικό για την κρίση, την ευελιξία ανάμεσα στους πυλώνες, το ανώτατο όριο και την εξωτερική σύγκληση. Ε, είναι ιδιαίτερα λυπηρό που το Συμβούλιο αρνήθηκε να ε, διαπραγματευτεί για αυτά τα ζητήματα, διότι είναι ζητήματα συναπόφασης και όχι πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό και ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να θεωρηθεί αυτός από απόπειρα του Συμβουλίου να αφαιρέσει ε, τις νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συναπόφαση. Ε, και λυπάμαι διότι οι Υπουργοί Γεωργίας ε, αρνήθηκαν ε, να ξεκινήσουν τη συζήτηση. Αυτό είναι ένα χτύπημα κατά της διαδικασίας συναπόφασης και της ίδιας της συνθήκης της Λισαβόνας. Ξέρουμε ότι κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα τελευταία δύο-τρία δύο, χρόνια έγιναν σοβαρές προσπάθειες και θα ήθελα να ποτίσω από ε, να απευθύνω εύσημα μάλλον σε όλο το επιτελείο μου και στη Γραμματεία των Συναρμοδίων Επιτρόπων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τζόρτζ. Ο Τζιμ Νίκολσαν τώρα. Τζιμ, Μάρτιν, έχετε το ίδιο peso, chi vuole. Είσαστε οι σοβαροί, ο Μάρτιν ή ο Τζιμ. Ο Μάρτιν, εντάξει. Ξεκινήσω. Και εγώ πρώτα μετά με τις ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στις συμβαστικές λύσεις και στις διαπραγματεύσεις βέβαια και από πλευράς του Κοινοβουλίου αλλά και από πλευράς ε, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, τον Επίτροπο και πάνω απ' όλα το, για το πολύ οικοδομητικό πνεύμα που είδαμε τελευταία εβδομάδα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Από τη Δευτέρα μετά το Λουξεμβούργο είδαμε ότι πήγαιναν τα πράγματα καλά και ότι μπορούσε να φέρει αποτελέσματα εν τέλει η Λισαβόνα αν την αξιοποιεί το Κοινοβούλιο. Εμεί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη στην ομάδα μου τη συζήτηση. Μπορώ να εκτιμήσω θετικά, αλλά με προσεκτικά θετικά τα αποτελέσματα αυτά ε, κυρίως με το πρασίνισμα. Κυρίως αν αξιοποιήσουμε τις λύσεις αυτές που μας δίνονται με το πρασίνισμα και στην πράξη πρέπει να κριθεί το πρασίνισμα τι είδου αποτέλεσμα φέρνει γιατί θέλουμε να μην είναι ένα greenwashing, ένα ξέπλυμα προς το πράσινο, αλλά ε, μια αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, μια αλλαγή υποδείγματος όπως λέμε. Και έτσι ε, και στις ε, πληρωμές 30% για το περιβάλλον στον πρώτο πυλώνα που θα πρέπει να αξιολογηθεί ως διαφοροποιημένα, γιατί εγώ μπορώ να πω ότι βεβαίως είναι μια επιτυχία όταν ε, έχουμε ένα 5% κατά προτεραιότητα πράσινες επιφάνειες και φτάνουμε στο 30%, βέβαια μπορεί να κρυθεί αυτό σε επιτυχία. Από την άλλη μπορεί να πει κανείς ότι στη διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν θα έχει καμία επίπτωση αυτό το πρασίνισμα, άρα θα έλεγα δεν αρκεί τις ε, πράσινες εκτάσεις ε, ε, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την προστασία του, του περιβάλλοντος, του κλίματος. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα κρίνουμε θετικά και μπορούν να σημάνουν αλλαγή συμπεριφοράς εφόσον υπάρχει επαρκής ανταπόδοση και οικονομική και άρα από εκεί θα κρυφθούν τα πάντα, δηλαδή αν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα μέτρα και γι' αυτό θέλω μεσοπρόθεσμα να υπάρχει η δυνατότητα της αξιολόγηση, αν ήταν αρκετά αποτελεσματική ή το πρασίνισμα, αποτελεσματικό το πρασίνισμα της γεωργικής οικονομίας στην Ευρώπη. Στη νέα κατανομή των μέσων δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στην εξωτερική και εσωτερική σύγκληση. Τα όσα έχουν προταθεί δεν αρκούν και μπορεί και στην προσεχή περίοδο να χρησιμοποιηθούν ε, για τις ε, πληρωμές στις ε, εκμεταλλεύσεις τα ιστορικά στοιχεία. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προχωρήσει γρηγορότερα. στη σύγκληση έχουμε προχωρήσει, πρέπει να το δουν αυτό τα κράτη-μέλη και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα σημαντικό βήμα προς την εξίσωση των ενισχύσεων. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα θετικό είναι ότι στις συνδεδεμένε ενισχύσεις το Κοινοβούλιο κράτησε και άντεξε με το 2% στις ε, συνδεδεμένες ενισχύσεις για την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ένα πρώτο βήμα ίσως αλλά πάντως ένα πολύ θετικό βήμα έτσι δεν εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τις αγωγές της σόγιας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταστήσουμε για όλα τα κράτη δεσμευτική την υποχρέωση ενίσχυσης των πιο αδύναμων, γιατί παραμένει στην επιλογή των, στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών η κατανομή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο των ενισχύσεων και η χορήγηση πιο σοβαρής ενίσχυσης προς το μικρό παραγωγό παρά στο μεγάλο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν ε, τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να δώσουν πιο δίκαιες ενισχύσεις στους μικρότερους παραγωγούς. Ε, εμείς ως Κοινοβούλιο Είχαμε προτείνει, ε, είχαμε ψηφίσει μάλιστα ένα νότατο επίπεδο, αλλά μετά μας είπε το Συμβούλιο ότι δεν έχουμε εντολή και δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα να συζητούμε τέτοιες ε, προτάσεις. Το κάπινγκ λοιπόν αυτό και για το πρασίνισμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά εάν τελικά πρόκειται να μην έχει και ένα αποτέλεσμα, ίσως ίσως είναι σκοπιμότερο να κοιτάξουμε τελικά μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή την πιο ισοδίκαιη κατανομή στις άμεσες ενισχύσεις. Για το δεύτερο πυλώνα συμφωνεί η ομάδα μου ότι τα αποτελέσματα για τη διαπραγμάτευση του δεύτερου πυλώνα θα τα υποστηρίξουμε και το 30% για το δεύτερο πυλώνα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα εκ μέρους της Ευρώπης ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά μέτρα για τη γεωργία. Και Ένα ζήτημα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι αν μπορούν μακροπρόθεσμα να παραμείνουν οι κατανομές των ποσών όπως έχουν μεταξύ του πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πιστεύω ότι τουλάχιστον δική μου την πατρίδα θα μείνουν οι πληρωμές όπως έχουν αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων από τους αρχηγούς ε, κυβερνήσεων ε, είναι πολύ δυσάρεστα. Είναι, πολύ, είναι απαράδεκτο για το Κοινοβούλιο να γίνονται εσωτερικέ διαβουλεύσεις και ε, παζάρια και τελικά να αποφασίζουν και να μας ανακοινώνουν μια-δύο εβδομάδες πριν μόλις ε, ποια είναι η κατανομή των ποσών. Για τον αμπελοϊνικό τομέα θα περιμέναμε περισσότερα, αλλά έστω μπορούμε να το δεχθούμε. Για το, για το γάλα όμως δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι, γιατί δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε μια σαφή ρύθμιση, μια ρύθμιση που να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Τα πολιτικά μέσα που είχαμε στα χέρια μας ε, για την ε, διαχείριση των κρίσεων μόνο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο όταν ξαναρχίσει με μια διάσκεψη τη συζήτηση του θέματος αυτού μπορεί να δώσει νέες προτάσεις και προοπτικές για τον ε, τομέα του γάλακτος. Λυπούμε που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να εξασφαλίσουμε περισσότερε πρόοδου στο σημείο αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν να καταλήξουν επιτυχώ οι συνομιλίε. Ένα άλλο θέμα για την εκθεσιλαβία εγώ ως πράσινος μπορώ να αισθάνομαι ικανοποιημένος για το ότι οι πληρωμέ και οι βασικέ ενισχύσει εν τέλει, το πρασίνισμα συγγνώμη και οι βασικέ ενισχύσει εν τέλει συνδέονται, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι σε εκούσια βάση το πρασίνισμα. Το βρίσκω πολύ θετικό αυτό και μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα, μπορούμε να δεχθούμε αυτή την πρόταση, όχι ολόκληρη την έκθεση, αλλά το συγκεκριμένο σημείο οπωσδήποτε. Άλλε ομάδε ίσω το ανέφεραν νωρίτερα, το επαναλαμβάνω και εγώ, ότι πάντα, τα πάντα τα συστούμε με την επιφύλαξη τη συμφωνία του μεσοπρόθεσμου ε, δημοσιονομικού πλαισίου Τίποτα άλλο δηλαδή δεν μπορεί να κριθεί πριν να κριθεί και αυτό, πριν να λήξει και αυτό. Και όσον αφορά την εντολή του Κοινοβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν πρόκειται να αφήσουμε να μας ε, ε, περιορίσει κανείς τη δυνατότητα των χειρισμών και την εντολή του Κοινοβουλίου. Ε, γι' αυτό έχουν μπει διάφορα πράγματα στις αγγίλες και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε την ε, τελική συμφωνία για το πολυεδρικές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα τα άλλα ήταν, ε, τα έχω καλύψει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Νίκολσον, έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως πρόκειται για την μεγαλύτερη διαπραγματευτική διαδικασία την οποία έχουμε δει και νομίζω ότι δεν, ε, δεν αισθάνονται ανακούφιση μονάχα η Γεωργία, αλλά νομίζω ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει να πω ότι η δικιά μου ομάδα δεν έχει ε, ακόμα αποφανθεί ποια θέση θα κρατήσει γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Επομένω έχουμε μια επιφύλαξη. Υπάρχουν πάντως ε, πολλά σημεία μπορούμε να, ε, με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οι άμεσες πληρωμές Πολλά πρέπει να γίνουν ε, και ενδεχομένως μπορώ να πω από τώρα ότι ε, ενιαία οργάνωση αγοράς ε, ενδεχομένως δεν θα μας βρει σύμφωνους. Αυτό το λέγαμε και από την αρχή άλλωστε. Η διαδικασία λοιπόν μας οδήγησε στο να ε, έρθουμε πολύ σε επαφή μαζί μεταξύ μας ε, και παρά τις διαφορετικές απόψεις ε, οδηγηθήκαμε στο σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον ακριβώς επειδή αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε πολύ μαζί και νομίζω ότι πολλά μάθαμε ο ένας από τον άλλον. Τέλος, προσωπικές σκέψεις ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου, εσένα προσωπικά ε, Σάιμον, αλλά και τον Επίτροπο ε, Τσιόλος ε, για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγαν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Να ευχαριστήσω το, τους διαπραγματευτές ε, γιατί ήταν πάντα διαθέσιμοι, ανοιχτοί, ευγενείς, καλοσυνάτοι ε, και ε, νομίζω ότι Σάιμον το να έχεις τέτοια καλά λόγια από μένα είναι μπόνους, έτσι πρέπει να το καταλάβεις αυτό, δεν, δεν το κάνω κάθε μέρα. Θα ήθελα βεβαίως και εγώ να ευχαριστήσω την δικιά μου ε, ομάδα. Ξέρετε, να μην ε, ξεχνάμε ότι οι μικρότερες ομάδες σε αυτό το κοινοβούλιο στρεσάρονται πολύ περισσότερο γιατί προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με πολύ λιγότερο ε, προσωπικό και δυνατότητες. Κοιτάξτε, εδώ σε αυτή τη διαπραγμάτευση ούτε χρόνο μετρήσαμε, ούτε οδηγίες για το χρόνο εργασίας ε, ε, σεβαστήκαμε, ούτε τίποτα. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω λοιπόν ε, τους πάντες. Βέβαια, το ερώτημα είναι, με όλη αυτή τη διαδικασία και όλο αυτόν τον κόπο θα βελτιωθεί η ζωή των γεωργών στην Ευρώπη και καταλήγω στο να απαντήσω όχι. Θα μειωθεί η γραφειοκρατία. Όχι. Θα ήταν ευκολότερο ε, οι γεωργοί με τη νέα διαδικασία να ε, διασφαλίσουν ε, την σωστή διαδικασία της αλυσίδας τροφίμων. Όχι. Πολλά θα ζητηθούν από τους γεωργούς, οι οποίοι τελικά θα πάρουν πολύ λιγότερα. Όμως τα πράγματα έχουν όπως έχουν, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. και το βέβαιο είναι ότι οι γεωργοί θα χρειαστούν μεγαλύτερη στήριξη ε, από την ίδια την αγορά έτσι ώστε να μην ε, στηρίζουν, αφού δεν θα στηρίζονται πλέον από την κοινή γεωργική πολιτική. Είμαι από την ε, Βόρεια Ιρλανδία όπως δυστυχώς μαρτυράει και η τρομερή μου προφορά. Να ευχαριστήσω ε, του την ε, ε, το Συμβούλιο για την καλή του στάση και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε και κάποια πιο ειδικά προβλήματα αυτής της συγκεκριμένης περιοχής. Επομένως, προσδοκώ σε αυτή τη συνεργασία. Λοιπόν, μερικές προσωπικές ε, ε, παρατηρήσεις. Πριν από 24 χρόνια ε, εξελέγει πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ένα μήνα δηλαδή θα κλείσουν τα 24 χρόνια. νομίζω ότι είμαι ο μακροβιότερος και παλαιότερος. Είδα και τις μεταρρυθμίσεις Μαξάρη και Φίσερ και όταν ήρθα εδώ είχαμε ένα σωρό ε, ε, προϊόντα σε καλές τιμές. Είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα. Ναι, περάσαμε από πολλά. Και να μην λησμονούμε ότι οποτεδήποτε είχαμε προβλήματα και οποτεδήποτε έχουμε προβλήματα στην κοινή γεωργική πολιτική ε, δεν πρέπει να λησμονούμε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση τώρα. Στο παρελθόν σε παρόμοιες περιστάσεις βλέπω ε, βουλευτές που δεν έχουν τίποτα να πούν και κοιτούν απ' έξω τη διαδικασία. Ενώ εδώ πραγματικά θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ θετικό βήμα προς το εμπρός. Για πρώτη φορά πιστεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σαν μέλη της Επιτροπής ε, ε, Γεωργίας μπορέσαμε να υψώσουμε τη φωνή μας, να ακουστεί η φωνή μας, να έχουμε input, να έχουμε δυνατότητα επιρροής για το τι θα συμβεί τα επόμενα 7-10 χρόνια. Ό,τι καν είναι αυτό. Ενδεχομένως κανείς μας δεν θα είναι απολύτως ευτυχής ε, ε, με, όλ, με τις αποφάσεις. Μερικοί θέλουν περισσότερο, άλλοι θέλουν λιγότερο, άλλοι λένε γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Όμως ε, έχω την εντύπωση ότι εδώ τούτη τη φορά η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είχε και το δικό μας το στίγμα. Τουλάχιστον είπα, εγώ μπορούσα να πω την άποψή μου. Έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου για αυτήν την ΚΑΠ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ευκαιρία για μας να προχωρήσουμε, να μάθουμε από τα κράτη-μέλη, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Και ε, ε, θα ε, ξέρουν όλοι ότι στην ιστορία της ΚΑΠ αυτή η απόφαση, αυτή η στιγμή ήταν μια στιγμή καμπής. Ευχαριστώ, Τζιμ, λέει ο Πρόεδρος δεν βλέπω τον, συντονιστό, ε, τον συντονιστή Άγνιου της Ευρώπης της Ελευθερίας και Δημοκρατίας, αλλά βλέπω έναν συναδελφό του, παρακαλώ αν θέλει να μιλήσει εξ ονόματος της ομάδας του. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για την εργασία που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πολύ μήνες αυτές οι διαπραγματεύσεις και πολλές οι απαραίτητες υποχωρήσεις και οι απαραίτητες συμβιβασμοί. Η διαπραγματευτική ομάδα λοιπόν αξίζει συγχαρητηρίων. Αναρωτήθηκα εάν η τελευταία, το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του Λουξεμβούργου ήταν απαραίτητο ή όχι ε, και αν οδήγησε σε καλύτερο αποτέλεσμα. Ε, με ενοχλεί λίγο που το λέω, αλλά νομίζω ότι δεν βοήθησε σε τίποτα το πρασίνισμα, το οποίο βεβαίως όλοι επιθυμούμε, θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί ε, με πιο αυθόρμητο τρόπο, πιο φυσιολογικό κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, ο κατάλογος των ε, παραγωγών ε, που μπορούν να έχουν συνδεδεμένες ενισχύσεις δεν μας ευχαριστεί το αποτέλεσμα. 13 Μαρτίου, στις 13 Μαρτίου εμείς ψηφίσαμε ε, για την κατάργηση του καταλόγου αυτού. Πολλά λάθη μπορεί να έγιναν τα τελευταία χρόνια στα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Το, ε, η γεωργική πολιτική θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις, σε επιλογές δηλαδή, ορισμένες επιλογές πρέπει να μένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών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 δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση λόγω ενός άρθρου ε, του, των ε, συνθήκων. Ε, πρέπει να έχουμε στο νου μας μόνο τους γεωργούς, την, τις ανάγκες που έχουν. Παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ένα βήμα ανάπτυξης και όπως έλεγε και ο συνάδελφος Νίκολσον, εδώ κάναμε ίσως ένα πρώτο κρίσιμο βήμα. Στο μέλλον θα πάμε ακόμα καλύτερα καλύτερα. Αυτό θα αποτελέσει βάση για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος ε, της ε, Γκουέ Ρούμπιξ. Και έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει με τους συντονιστές όλων των ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Μπορώ να συμφωνήσω στο μεγαλύτερο τμήμα των όσων είπαν οι συνάδελφοι. Έχουμε συζητήσει πολύ. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που είναι εφικτό το πράττουμε, αυτό που δεν είναι εφικτό το αφήνουμε. Πολλέ είναι οι συμβαστικέ λύσει που έχουν βρεθεί. Με κάποιε είμαι πιο ικανοποιημένο, με κάποιε άλλε λιγότερο. Φαίνεται να χαιρετίζουμε κάποια μεγάλη νίκη. Απαγγέλλονται μεγάλε ομιλίε και λόγοι. Αλλά το τι τελικά έχουμε επιτύχει, ο Γεωργό τη Ευρώπη θα το αξιολογήσει και θα το εκτιμήσει. Και μπορεί ίσω αυτό να μην δείξει τόσο πολύ ενθουσιασμό όσο εμεί σήμερα. Αλλά το να βρεθεί συμβασμός δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα τον ακολουθήσουν τον συμβασμό όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό. Εμείς πάντως και η ομάδα μου μπορούμε να υποστηρίξουμε την κατεύθυνση που έχει επιλογή, επιλογή που ακολουθεί αυτός ο ε, συμβασμός για τις άμεσες ενισχύσεις βλέπουμε ακόμη να παραμένουν κάποιες ανισότητες για τους πιο νέους αλλά και τους πιο ηλικιωμένους γεωργούς. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και ανάγκη για ενίσχυση. Δεν θέλω να επαναλάβω τις θέσεις μου. Ιδιαίτερα ε, τρέφω εκτίμηση για τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τα θέματα όλοι οι εμπλεκόμενοι στις ε, οι εμπλακέντες της διαπραγματεύσεις ε, και ο κύριος Δεκάστρο και ο κύριος ε, Επίτροπος και εγώ έλαβα ένα, σε ένα βαθμό μέρος διαπραγματεύσεις και διαπιστώσα προσωπικά πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των εισηγητών. Ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας στο βαθμό που μπορούμε και ελπίζω και εύχομαι για τους πάντες, για όλους μας εδώ αλλά και για τους γεωργούς της Ευρώπης στο μέλλον να εφαρμοστεί πραγματικά και στην πράξη αυτός ο συμβασμός, αυτή η λύση, γιατί εάν δεν υλοποιηθεί, αν δεν εφαρμοστεί πραγματικά, ό,τι και να συζητάμε εδώ, είτε για 40 μιλάμε, είτε για 50, είτε για 60 τριμερείς διαλόγους και για τέρμονες ώρες όπου θα αναζητούνται λύσεις, δεν θα έχουμε φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η ιστορία θα δείξει αν ήταν δηλαδή καλή επιλογή. Με, από την εφαρμογή θα κρυθεί. Ας περιμένουμε λοιπόν και ας δούμε. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και γυρνάω στον ε, γύρο των, ε, των συντονιστών. Βλέπω ότι υπάρχει γενικότερα συμφωνία για, την, ε, για να υποστηριχθεί αυτή η συμβαστική πρόταση. Τώρα κοιτάμε τους, ακούμε τους όδης συγκητές και όλους τους συναδέλφους που έχουν στο λόγο και παρακαλώ να σεβαστε όλοι τους χρόνους ομιλίας. Έχουμε ένα χρόνο περίπου ούτε καν μία, 50 ε, λεπτά, ούτε καν μία ώρα, ε, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε τις συνεδρίες, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου όπως είπαμε. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε πόσο χρόνο αγόρευση έχω στη διάθεσή μου. Ε, πάλι να κάνουμε διαπραγματεύσεις, να κάνουμε συμφωνία. Λοιπόν, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Πολλοί θεωρούν, παραδείγματο χάρη οι ακροατές μας πίσω-πίσω ε, στην αίθουσα, να πιστεύουν ότι ήταν όλα ρόδινα όπω και το αποτέλεσμα. Όχι, ήταν όλα πάρα πολύ σκληρά, σκληρές διαπραγματεύσεις ε, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή, ο επίτροπο ε, χαμογελάει τώρα, αλλά υπήρχαν, υπήρξαν πολλέ στιγμές που δεν χαμογελούσαμε καθόλου. και, η πολιτική, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επιτελείο μας ε, το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Θα θέλαμε λοιπόν να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους όσους εργάζονται χωρίς να φαίνονται και πρέπει να τους αποδοθούν εύσημα. Να σας πω ε, και κάτι που διαφέρει από την προηγούμενη μεταρρυθμιστική πολιτική, το Twitter. Έτσι μπορούμε να έχουμε τις απόψεις ε, όλων στιγμιαία. Παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο μπόρεσε να αποφανθεί εγκαίρως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μας είπε κινδυνεύει το περιβάλλον εξαιτίας της Γεωργικής Συμφωνίας. Όμως αυτό δεν αληθεύει, δεν ευσταθεί. Είχαμε πάντοτε κατά νου τις επιπτώσεις για το περιβάλλον. 30% των πληρωμών προς τους γεωργούς συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα στον περιβαλλοντικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να προβληματιστούν και να δουν τι θα γίνει και γι' αυτό έχουμε προβλέψει ενδιάμεση αναθεώρηση για τη νέα πολιτική. Πρόκειται για μεγάλη καμπή. Το είπατε στην εναρκτήρια ομιλία σας. Ε, το πρασίνισμα ε, σηματοδοτεί μια νέα εποχή και ε, κατοχυρώνει την προστασία του περιβάλλοντος ενώ κατοχυρώνται και τα εισοδήματα των γεωργών. Η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι στον πυρήνα της προσπάθειας μας. Θέλω να το τονίσω. Οι γεωργοί δε είναι ενθουσιασμένοι διότι εμείς αγωνιστήκαμε για το υποχρεωτικό σύστημα εναντίον τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την συνολική πληρωμή, για το συνολικό ποσό της πληρωμής. Ε, επίσης ενθαρρύνουμε τους νέους γεωργούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, σε σχέση τώρα με τη συνολική συμφωνία για τις ε, άμεσες πληρωμές, ας είμαστε ειλικρινείς, ε, του ζητούμε να κάνουν περισσότερα με λιγότερα μέσα, οπότε θα πρέπει να δούνε από πού θα πάρουν το εισόδημά τους, από την αγορά και από τις άμεσες ενισχύσεις. Νομίζω ότι εκεί δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, θα επανέλθουμε το φθινόπωρο. Δεν ξέρω η αγορά τι μέρος του εισόδηματος μπορεί να κατοχυρώσει για τους γεωργούς για τη διαδικασία συναπόφασης. Ε, και όντως μάθαμε όλοι πάρα πολλά. Ε, ε, έχουμε αντλήσει διάφορα διδάγματα από όλη τη διαδικασία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Πάντως ήταν πάρα πολύ θετικές οι εξελίξεις. Εγώ συζήτησα με Ιρλανδούς γεωργούς και άλλους σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διαβεβαίωσαν ότι είναι ικανοποιητική η συμφωνία. Θα γίνουν αλλαγές και προσαρμογές για πολλούς γεωργούς και πρέπει να τους δώσουμε χρόνο για να τα καταφέρουν αυτό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ακριβώς ακριβώς αυτό το ρόλο να συνοδεύσουμε τους γεωργούς. Είναι ακέραιοι όμως οι γεωργική μας πολιτική. Έχουμε το κονδύλι, είναι βιώσιμοι ε, και έχουμε αυτά αποτελέσματα για τους γεωργούς, για τους πολίτες και για το περιβάλλον. Ε, ας υποκληθούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Γκαρσία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ, ως ήθιστε, και όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ε, θα ξεκινήσω λοιπόν ε, ευχαριστώντας ε, τους βοηθούς μας, τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, τους συγητές, Μισελ Νταντάμ, τον οποίο είχα την τύχη να δουλέψω στα πλαίσια του θέματος της κοινής οργάνωσης της αγοράς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον σύντροφο ε, ε, Καπόλας Σάντος γιατί ξέρω ότι αναγκάστηκε να σχηνοβατήσει έτσι ώστε να ε, μπορέσει να βρει ε, λύσεις που να ικανοποιούν ε, πολλούς και να είναι ισορροπημένες. Ξέρουμε ότι έπρεπε να γίνουν βελτιώσεις, αλλά εδώ μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Βεβαίως, το τελικό αποτέλεσμα αυτού του τριμερούς διαλόγου, αυτής της πολιτικής συμφωνίας, είναι ένα συν. Τώρα, η συμφωνία θα μειώσει, θα αμβλύνει ε, τις αρνητικές επιπτώσεις ε, σε κάποιους τομείς που οπωσδήποτε θα φυγούν, το βέβαιο είναι πως ναι. Αλλά μην λησμονούμε ότι παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν ε, θα υπάρξουν κάποιοι τομείς εκτινοτροφίας και γεωργίας που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες η υλοποίηση ε, αυτής της συμφωνίας ε, θα είναι ευαίσθητη για κάποιους τομείς και επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε εν τέλει ε, να μην εκλείψει η κτηνοτροφία και η γεωργία. Το μέλλον της υπαίθρου στην Ευρώπη εξαρτάται από τις συμφωνίες αυτές. Ε, είναι ένα επικίνδυνο εντό εισαγωγικών ε, μέλλον. Ε, βεβαίως πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, πρέπει να λύσουμε και τα προβλήματα που εξακολουθούν να παραμένουν. Θα τελειώσω με τα δημοσιονομικά ζητήματα. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Τούτη η συμφωνία δεν θα μπορέσει να ψηφιστεί όσο δεν γνωρίζουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπενθυμίζω τις απαιτήσεις μας, ε, Σάιμον, ε, τις ανάγκες μας. Ε, πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να δεχτεί αυτή την συμφωνία. Το πει. πρέπει να ψηφιστεί γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ούτε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Πρίτα Ρέμις και μετά Κόστιντζερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως και το θέμα της ε, προστασίας ε, της εργασίας που έχει παραμεληθεί. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Νταντάιν που πάντα έδειξε καλή διάθεση να ακούσει, να αποδεχθεί προτάσεις, να τη συζητήσει ακόμα και αν δεν είχαμε πάντοτε την ίδια θέση, αλλά αυτό βέβαια είναι, μέσα, είναι κομμάτι της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Θέλω να ευχαριστώ μετά τους διερμηνείς, λέει η κυρία Κόσιγκερ, γιατί χρειάστηκε να εξοικειωθούν με τόσο περίπλοκους ε, όρους ε, και έννοιες εδώ με τη γεωργική πολιτική που ξέρω ότι δυσκόλεψαν πολύ. Και θα θυμίσω το ρητό το καλό πράγμα αργεί να γίνει χρειάστηκε να δώσουμε χρόνο να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε από πολύ διαφορετικές τοποθετήσεις και θέσεις και παρόλα αυτά καταφέρνουμε νομίζω έστω και με την πίεση αυτού του χρόνου που είχαμε προς το τέλος να ολοκληρώσουμε Ίσως να μην είμαστε όλοι απολύτως εκατονοποιημένοι, ίσως κάποιοι να πιστεύουμε ότι δεν ήταν όλα τέλεια και ότι δεν τα καταφέραμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε ή όσο θα μπορούσαμε. Αυτό αποτελεί και ένα μάθημα, ότι μπορούμε να δαχθούμε για το μέλλον, ε, να προχωρούμε ίσως πιο γρήγορα με τη δουλειά μας, στη δυνατότητα της συνεργασίας και των ε, ε, διαπραγματεύσεων. Εμείς μαζί με τους συνεργάτες μας έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι και στο μέλλον μπορούμε πιο συστηματικά να εργαζόμαστε και πιο, σε πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων να προχωρούμε και να πλησιάζουμε ένα θέση του άλλου. Η ομάδα μας την εβδομάδα αυτή δεν είναι παρούσα στις Βρυξέλλες. Έχουμε ένα εξωτερικό, μια εξωτερική εκδήλωση της ομάδας, έξω από τις Βρυξέλλες δηλαδή, και έτσι δεν μπορούμε να εκδηλώσουμε ε, θέση ως ομάδα στο Στρασβούργο με την ησυχία μας ήρεμα ήρεμα θα καταθέσουμε απόψεις και θέσεις και θα δώσουμε μια ετοιμιγορία. Ε, πάντως εκ του προχείρου μπορώ να πω ότι σαν να ξυπνήσαμε όλοι από μια χειμερή ανάρκη ξαφνικά. Ίσως ξαφνικά αρχίζουμε να συναισθανόμαστε ότι ήρθε το καλοκαίρι και ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Αλλά είμαστε και όλοι πολύ κουρασμένοι. Αποδείξαμε πάντως ότι έχουμε τη δύναμη να δώσουμε όλη μας την ενεργητικότητα σε μια προσπάθεια μεγάλη και να φέρουμε αποτελέσματα. Πρόκειται για μια καλή συμβαστική λύση για την Ευρώπη και όπως και να έχει θα δούμε και θα κριθεί αυτή η συμβαστική λύση, ε, η επιτυχία της, από την εκτέλεσή της στην πράξη. Θα δούμε και στα κράτη που έχουν ομοσπονδιακές δομές όπως η Γερμανία το πώς θα υλοποιηθεί στα επιμέρους κρατήδια, γιατί δεν έχουμε μόνο μια κεντρική διοίκηση να αντιμετωπίσουμε, αλλά και τα επιμέρους κρατήδια. Και ξέρετε ότι πολλές φορές αυτό μπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. είσαι αποτελέσματα λοιπόν βλέπουμε συχνά ως προς την ε, υλοποίηση από πλευράς της διοίκησης, της γραφειοκρατίας ε, λύσεις οι οποίες μπορεί σε κάποιο άλλο κρατήδιο ή κράτος να φαίνονται πολύ πιο ικανοποιητικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόστιγκερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας το προσωπικό του δικού μου γραφείου, αλλά βέβαια και της ομάδας για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει στη διαδικασία αυτή της συναπόφασης και μας υποστήριξαν μέχρι τέλους. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί προχωρήσαμε με πολύ δύσκολα βήματα, αργά βήματα ε, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και, τα προγράμματα οικολογικά καταφέραμε να μην περικοπούν πάρα πολύ πράγμα το οποίο αποτελούσε ένα σοβαρό κίνδυνο γενικά για την κοινή πολιτική να μην δούμε μια πραγματική και καλή μεταρρύθμιση. Ένα καλό βήμα λοιπόν, για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι εν τέλει. Τώρα το πόσο εφικτή θα είναι η εφαρμογή του στην πράξη, πόσο πρακτικά εύκολη θα είναι η υλοποίησή του, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Δεν απλουστέψαμε πάντω τη γεωργική πολιτική. Αυτό δεν το καταφέραμε. Χρειάστηκε σήμερα να εξηγήσω το μοντέλο της, ε, ε, των ισοδυνάμων και για την ομάδα μου. Δεν είναι εύκολο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι έχουν γίνει πολλές μεγάλες προσπάθειες. Και δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο το αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε καταλήξει. Οι καταναλωτές αλλά και ο Γεωργός της Ευρώπης απαιτεί, περιμένει από εμά για, για την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, λύσεις οι οποίες καταγράφονται βέβαια σε αυτά τα άρθρα, αλλά ταυτόχρονα θα εξαρτηθεί η επιτυχία τους από την τελική υλοποίηση. Οι αρχηγοί λοιπόν κρατών και κυβερνήσεων που έχουν και να ε, καταλήξουν ακόμη σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, σε ένα δημοσιονομικό, ε, στους δημοσιονομικούς πόρους, θα πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε να μην εξουδετερώσουν τα καλά αποτελέσματα αυτής της ε, πρότασης. Για τη γραφειοκρατία, σε ένα βαθμό έχουμε μπορέσει να απλουστεύσουμε τις προτάσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και το θέμα του νέου γεωργού, του πρώτο ε, απασχολούμενου στη γεωργία. Έχουμε κάποιες καλές λύσεις, πιστεύω, εξασφαλίσει για τους γεωργούς μας που μπορούμε στο μέλλον να τους βοηθούμε. Για την ασφάλιση κινδύνου και το μέσο σταθερότητας, το μόνο που μπορώ να πω είναι να φέρει αποτελέσματα και για το μέλλον, γιατί έχουμε, πατήσει, έχουμε βρεθεί σε νέο έδαφος, ε, αχαρτογράφητη περιοχή και πιστεύω θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση σε επίπεδο κρατών μελών και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια να την παρακολουθεί πολύ προσεκτικά ώστε να ε, στεφθεί με επιτυχία για το μέλλον. Για τις ε, περιοχές που έχουν ε, δυσμενείς συνθήκες, που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε. Είναι πολύ ευαίσθητες οι περιοχές και αν δεν δώσουμε σε αυτές ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή, θα έχουμε ειστερήσει σε σχέση με μια μεγάλη ευρωπαϊκή ευθύνη. Πρέπει λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή, αναλογικότητα και ε, συνείδηση της σημασίας τους να φροντίσουμε αυτές τις μειονεκτικές περιοχές. Για τον τομέα δε των ορεινών, των ορεινών περιοχών ιδιαίτερος, θα ήθελα να επισημάνω ότι ιδιαίτερη σημασία είχε να μην θεσπιστούν ανώτατα όρια για τον τομέα των ορεινών περιοχών. Θέλουμε να έχουμε βεβαίως ε, την εκτατική αυτή γεωργία στις ε, κάτω, στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και μια ανάπτυξη της υπαίθρου εκτεταμένη. Ποιότητα λοιπόν ζωής, ιδιαίτερα χάρη στην ανάπτυξη της υπαίθρου για κάθε περιοχή της Ευρώπης και πιστεύω ότι εδώ πλέον, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ποσοστά της χρηματοδότησης, μπορούμε να βρούμε στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου τα κατάλληλα ποσά για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους και ιδιαίτερα ε, όλους τους συγητές που επέδειξαν τόση ε, ε, υπομονή έναντι μου όπως άλλωστε και όλοι οι συνάδελφοι στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ Λίσοκ και Κανιέτε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους συναδέλφους πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαβία και μετά τους υπόλοιπους εισηγητές, αλλά φυσικά και όλο το staff το οποίο ε, μας ε, στήριξε και να ευχαριστήσω ε, και όλους τους υπαλλήλους και του Συμβουλίου και της Κομισιόν που μας βοήθησαν με υλικό, με γραφήματα, με πίνακες κτλ. Κοιτάξτε, κάθε μεταρρύθμιση έχει ένα κόστος. Εδώ έχουμε μία ανοιχτή μεταρρύθμιση που ανοίγει δρόμους δηλαδή, που μας δίνει πολλές δυνατότητες. Όσον αφορά το greening, αυτά είναι προγράμματα τα οποία εάν υλοποιηθούν σωστά καθόλου δεν θα ζημιώσουν τους γεωργούς ε, του Ναντίον. Θα είναι και πάρα πολύ καλά για το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλες αυτές τις φωνές που λένε ότι δεν θα υπάρξει απλούστευση της ε, ΚΑΠ. Βεβαίως θα υπάρξει απλούστευση και μέσα από αυτές τις οριζόντιες ε, λύσεις της ΚΑΠ μπορούμε να φτάσουμε σε πολυετείς συμφωνίες οι οποίες πολύ μειώνουν και το διοικητικό και το οικονομικό κόστος. Έχουμε επίσης μέτρα για την ε, παροχή συμβουλών στους ε, ε, γεωργούς και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Επίσης, όσον αφορά τον υπολογισμό των λαθών που μπορεί να προκύψουν ε, στη συμπλήρωση των αιτήσεων ή των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ. Ε, έχουμε λάβει μέτρα έτσι ώστε να γίνονται οι έλεγχοι, να είναι αποτελεσματικοί, αλλά να μην είναι κυρωτικοί από την πρώτη στιγμή για τους γεωργούς. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια ε, σημεία επί των οποίων δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε επιβεβαίωση της θέσης μας. Ξέρετε, ε, όλοι οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουν τις ίδιες άμεσες ενισχύσεις. Ε, είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο τα νέα κράτη-μέλη αλλά και τα παλαιά. Ελπίζω ότι στο μέλλον ε, θα αλλάξουν αυτά. Επίσης να πω ότι υπήρξαν και μειώσεις όσον αφορά την χώρα μου, την Πολωνία ε, κατά 26% για τα γεωργικά περιβαλλοντικά προγράμματα, για τους νέους ε, γεωργούς, ε, για τις γυναίκες στην Ήπεθρο, προγράμματα σε σχέση με τον εξυγχρονισμό κτλ. Μεγάλη μείωση από το δεύτερο πυλώνα και αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ έχουμε δηλαδή μείωση κατά το 1 τέταρτο για την ε, ε, ε, γεωργία στην Πολωνία και αυτό ισχύει και για άλλες χώρες μέλη και μάλιστα σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι υποχρεωμένη πλέον αλλά έχει και τη διάθεση να συνεργαστεί με τις ε, ε, χώρες μέλη. Τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν με τρόπο τέτοιο ώστε οι στόχοι για τους οποίους πολλής λόγος έχει γίνει να επιτευχθούν. Αύξηση της γεωργικής παραγωγής, αύξηση των, των τροφίμων στην Ευρώπη, προστασία του περιβάλλοντος ε, και άνοιγμα δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ε, Ήπεθρο. Αυτές είναι, αυτή είναι η στόχη. Και επίσης αναφερόμαστε και στην αύξηση της ε, ποιότητας. Ο ρόλος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ. Σάντρα Κανιέτε και μετά Έκνουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ηγητές και τους σκιώδεις ηγητές καθώς και το προσωπικό για ε, τη σκληρή δουλειά τους και την ενέργεια που επένδυσαν στη διαδικασία. Είχα την τύχη να μετάσχω κι εγώ στη διαδικασία και να επηρεάζω και τις εξελίξεις μάλιστα για τις ε, άμεσες πληρωμές, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους γεωργούς στις βαλτικές χώρες. Θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα προς τον Υπουργό και προς τον Επίτροπο. Τι θα συμβεί στο μέλλον ε, όταν τα τρία ζητήματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν διότι εντάσσονται στο, στις διαπραγματεύσεις του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ποιος θα λάβει τις αποφάσεις, ποιος θα λάβει τις αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο του Πουδουπού, διότι βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας προκύπτει ότι αποκλείεται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων το Κοινοβούλιο δεν θέλουμε να δημιουργηθεί ε, νομικό προηγούμενο κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, το ίδιο ισχύει και για την εντολή που είχαμε για την εξωτερική σύγκληση. Ευχαριστούμε, Σάντρα. Παρακαλώ πολύ να μην ξεπερνάτε τον ε, χρόνο σας. Η Σάντρα ήταν σύντομη και αποτελεσματική. Thank you, Mr. Uh, ευχαριστώ. Θα αρχίσω με τον ε, οριζόντιο κανονισμό, διότι εγώ ήμουν ε, σκιώδης για τους ε, πράσινους και ευχαριστώ τον κύριο Λαβία. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας. Ξέρετε ότι εμείς το Μάρτιο καταψηφίσαμε τον κανονισμό Βλέπουμε τώρα όμως αλλαγές και βελτιώσεις από τη δική μας οπτική γωνία, κυρίως όταν μιλάμε για τους συμβουλευτικούς μηχανισμούς για τους γεωργούς και την επιβολή κυρώσεων που υπερβαίνει το 30% του πρασινίσματος. Πολύ σημαντικά σημεία για μας και ε, φυσικά χρειάζεται ε, πιο εκτεταμένη συζήτηση, αλλά ενδέχεται να αλλάξουμε ε, τη θέση που έχουμε υιοθετήσει και να υπερψηφίσουμε. Όμως χρειαζόμαστε πολιτική δήλωση για την οδηγία για τα παρασιτοκτόνα και θέλουμε να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σημειωθεί η πρόοδος. Επίσης, φυσικά το θέμα των άμεσων πληρωμών για το ανώτατο όριο, το κάπινγκ, είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Όταν δω, βλέπουμε το πρασίνισμα, οι πράσινοι θεωρούν ότι δύο είναι τα βασικά ζητήματα. Πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα που συμφωνήσαμε για το πραγματικό πρασίνισμα. Πολύ ωραία να διατύπωση, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Αυτό δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο και δεν είμαστε πεπισμένοι ακόμη. Επίσης, ε, ε, ποια διαφορά με την καθεστική ατάξη, για να ε, τη συνειδητοποιήσουμε αυτό έχει σημασία για τους για τις άμεσες πληρωμές πρέπει να ε, καταλάβουμε τι ισχύει πρωτού αλλάξουμε τη θέση μας ε, για τις άμεσες ε, ενισχύσεις. Θα είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί διότι στο κάτω-κάτω της γραφής το πρασίνισμα πέρα από μια νέα λέξη στην κοινοτική ζαργόν θα πρέπει να σημάνει αλλαγή στην κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστούμε ο Ζωζέ Μποβέ και μετά Μάτο. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που ο εκπρόσωπος ε, του Συμβουλίου αποχώρησε τη στιγμή που παρεμβαίνω. Ίσως να επανέλθει, ίσως και να τα μεταφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι είμαι στεναχωρημένος. Στεναχωρημένος ε, εξαιτίας ε, των εξελίξεων στο φάκελο από τότε που ε, παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Τσιόλος. Αυτό το σχέδιο έχει αποσυνδεθεί στα εξών συνετέθη, αν θέλετε τη γνώμη μου. Υπήρξε μια νέα πνοή το 2011, αλλά έχει εκπνεύσει τώρα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με συγκεκριμένα μέτρα και επιμέρους σημεία. Θέλω να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το 2013... Το 2003 ε, η κυρία Φίσερ Μπολ πήρε μία σκούπα και τα πήρε και τα σήκωσε όλα στην κοινή γεωργική πολιτική μεταρρύθμιση πλήρης. Σήμερα το σημερινό σχέδιο ε, δεν οφείλεται σε λάθος ε, ούτε της Επιτροπής ούτε του Κοινοβουλίου. Είναι του Συμβουλίου. Δηλαδή επανεθνικοποιούμε αυτή τη στιγμή τις ε, εθνικές, τη γεωργική πολιτική και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το επανεθνικοποιούμε. Ιδού το πρόβλημα. Είτε μιλάμε για το ανώτατο όριο για την φθήνουσα αναπροσαρμογή, για το πρασίνισμα. Δεν έχει σημασία τι αποφασίζουμε, διότι δεν υπάρχει γενική κατεύθυνση. Και βλέπουμε λοιπόν, όταν εξετάζουμε τα μέτρα, ότι ε, το ανώτατο όριο δεν είναι ικανοποιητικό και το πρασίνισμα ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα γιατί οι μονοκαλλιέργειες μπορούν να συνεχιστούν ε, στο 90% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Γι' αυτό και θλίβομαι και λυπάμαι διότι ο Μισελ Νταντά ε, προσπάθησε να επιτύχει καλά αποτελέσματα για το φάκελο της κοινή ΚΟΑ, αλλά σήμερα το πρωί μας έδωσε το τελικό πλήγμα το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 43.3. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για οικονομικές αποφάσεις ε, θεμελιώδους σημασίας ε, ε, και μας απείλησε το Συμβούλιο. Είπε αν χρησιμοποιηθεί το 43-3 ως νομική βάση θα τα αρνηθούμε όλα. Είναι απαράδεκτη αυτή η απειλή και επίσης απαράδεκτο είναι τα κράτη-μέλη να αρνούνται μια ισότιμη μεταχείριση στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μεταξύ. Κέρδισε ε, με τον κόπο του τη θέση του στον τριμερή διάλογο το Κοινοβούλιο, όμως συνεχίζει το Συμβούλιο. Θέλει να περιθωροποιεί το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Ζωζέ. Μάτων Τροβέρ και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, ο, κόσμος έτσι πάει. Άλλος χαίρεται, άλλος λυπάται. Ο κύριος Μποβέ λυπάται, εγώ όμως ε, χαίρομαι. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο, Επίτροπε, τον κύριο Επίτροπο και τον Προεδρεύον του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο Δεκάστρο. Νομίζω ότι ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από μερικές εβδομάδες ε, αισθάνθηκα μεγάλη ικανοποίηση και πιστεύω ότι είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη. Προσπαθήσαμε πολύ, περάσαμε από δύσβατους δρόμους, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και νομίζω ότι βρήκαμε τον τρόπο να υπεραμεινθούμε ε, των ε, ε, κύριων αρχών της κοινής γεωργικής πολιτικής. Πιστεύω ότι κερδίσαμε τη θέση μας σαν κοινοβούλιο και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Ε, επεδείχθη η ευελιξία και αυτό επίσης είναι πολύ θετικό. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να σεβαστούν ε, τους ε, περιβαλλοντικούς κανόνες, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκομίσουν και αυτοί τα ωφέλη του πρασινίσματος. Η ενίσχυση ε, επιφάνεια ε, έδωσε τη δυνατότητα να μην μειωθούν δραματικά ε, οι επιδοτήσεις. Φτάσαμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Πρόεδρος, συνεχίζουμε με την κυρία Ντότσε και μετά ο Σένφος Ντίρλινγκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες για τη δουλειά σας αυτή τη διαδικασία της μεταρρύθμισης, αλλά και για τον Επίτροπο Τσόλος και τον ε, Υπουργό Κόβνη σε αυτή τη διαδικασία. Η Προστερή Γεωργή στη Βόρεια Ιρλανδία, την ε, εκλογική μου περιφέρεια, ενώ αντιμετωπίζουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δύσκολες αγορές. Πάνω απ' όλα θέλουν να γνωρίσουν ότι υπάρχει σαφήνεια, σαφές πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια, για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Και φαντάζομαι ότι όλοι σήμερα ρίξαν μια ματιά στο πρόγραμμα της Επιτροπής μας, περιμένοντας να δούνε τι είδους ε, συμφωνία προκύπτει. Μια συμφωνία μερική, πρέπει να πούμε, διότι τα σημαντικά στοιχεία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν, μπορούν να τα, δεν μπορεί να τα συστήσει το Κοινοβούλιο και ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί. Άρα δεν είναι σε φύση κατάσταση για τα επόμενα χρόνια. Οι υποστήριοι γεωργοί στη Βόρεια Ιρλανδία ζητούν απλούστευση της γραφειοκρατίας, του γραφειοκρατικού φόρτου με τον οποίο είναι αντιμέτωποι. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν τους βοηθάει. Και είναι πιο εκτεθειμένοι σε κυρώσεις από ό,τι ποτέ στο παρελθόν νομίζω. Η γεωργία είναι κλειδί για την οικονομία της Βόρειας Ιρλανδίας. Έχουμε περάσει στην οικονομία μας μια περίοδο πολύ δύσκολη. Έχουμε χάσει τέσσερις εργασίες. συρρυκνούται η οικονομία. Μια κοινωνική λοιπόν γεωργική οικονομία η οποία προάγει βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα είναι και κλειδί κέρια σημασία για τη λειτουργία της οικονομίας μας. Είναι ευπρόσδεκτη λοιπόν η συμφωνία, αλλά ανησυχώ ιδιαίτερως για το ζήτημα του ενεργού γεωργού και τις σχέσεις που θα έχει με τα δικά μας συστήματα στην Βόρεια Ιρλανδία. Ξέρω ότι έχουμε ένα πολύ περιορισμένο ορετικό κατάλογο σε σχέση με τον ενεργό γεωργό. Δεν αρκεί όμως αυτός, ώστε να εξασφαλίσουμε πως τα λεφτά θα πηγαίνουν σε αυτούς που παίρνουν λίγα λεφτά και τα λεφτά θα τα βάζουν στην παραγωγή καλών τροφίμων για τον φορολογούμενο. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη διαφάνεια, εδώ περισσότερη σαφήνεια. Ιδιαίτερα καλωσορίζω το μήνυμα για τον νέο Γεωργό. Την ιδέα, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί στην πράξη, ε, την ιδέα της περιφερειοποίησης της κυριαζιολικής πολιτικής και αναφέρθηκε η ειδική σημασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της άμεσης ανταπόκρισης. Η Επιτροπή σήμερα μας είπε ουσιαστικά ότι στην ε, Βρετανία, τη Σκοτία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Ουαλία. Ε, οι αρχές μπορούν να ορίσουν ένα το, όριο διαφορετικό ανάλογα με τις ε, προδιαγραφές και ανάγκες τους. Εγώ νομίζω ότι δεν θα χρειάζεται στο μέλλον αυτό να συμβεί με πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον ε, το γαλακτοκομικό τομέα που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τη γεωργία αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας στη Βόρεια Ιρλανδία είναι περίπλοκη κατάσταση, το ξέρω, αλλά όταν έχουμε απορρίθμιση των ποσοστώσεων και κατάργησή του το 2015, το να δίνεται ως μόνη απάντηση για τη γεωργική πολιτική ένα, μια υψηλού επίπεδου συνδιάσκεψη εφέτος, προφανώς δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, ε, χρειαζόμαστε πραγματικά εργαλεία παρέμβαση στην αγορά, εργαλεία που να είναι χρήσιμα, που να είναι αξιοποιήσιμα και τα οποία θα μας επιτρέψουν να ξανακοιτάξουμε την ε, τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2007-2009. Ξέρετε ότι οι παραγωγοί δεν ασχολούνται ούτε με τι διαπραγματεύσει ούτε με του κόπου μα και τα ξενύχια εδώ στι Βρυξέλλε. Θέλουν ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Θέλουν νομοθεσία που να του επιτρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Το πώ αισθάνονται σήμερα ίσω είναι πρόημο να το πω. Αλλά εγώ περιμένω να δω την πραγματική υλοποίηση του προγράμματο και καθώ προχωρούμε προ μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια, την ολοκλήρωση τη νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Γκέρλινγκ και μετά Γέγκλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία Γιέγλε πρώτα. Η κυρία Γκέρλινγκ πρώτα. Καλωσορίζω και εγώ όπως και όλοι οι υπόλοιποι τη συμφωνία γιατί ήταν βασανιστική διαδικασία και επιτέλους τελείωσε. Ο υπουργό Κόβενη όμως είπε στην αρχή ότι ε, θεωρεί ότι ότι επικρατεί μεγάλη ασφάλεια. Μα πού είναι, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πολλά ακόμη δεν έχουν συμφωνηθεί και αναμένουμε. Ε, ε, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να πάω τώρα στο κράτος μέλος μου και να εξηγήσω στους γεωργούς τι συνέβη. Ε, διότι ε, το σίγουρο είναι ότι θα χάσουν 30% από την πρώτη μέρα κιόλας ε, των πληρωμών, εκτός και αν εφαρμόσουν μέτρα πρασινίσματος που ενδείκνεται ή και όχι για τις ανάγκες της εκμετάλλευσής τους. Και θα χάσουν κι άλλα 30% εάν δεν συμμορφωθούν στη συνέχεια. Ε, μιλάμε για τα περιβαλλοντικά μέτρα και την εσωλορθή χρήση του πυλώνα 2. Αναρωτιόμαστε όμως σε χώρες όπως η δική μου από πού θα προέλθει η υποστήριξη. Γράφεται κάτω-κάτω στον πίνακα για τον πυλώνα 2 πράγματα που δείχνουν ότι το μέλλον δεν είναι τόσο ροδινό, συγγνώμη, για το περιβάλλον όπως μας τα περιγράφετε εσείς. Για την κοινή ΚΟΑ έχουμε την παρέμβαση, συνδεδεμένε συνδεδεμένες ενισχύσεις, είναι μακρύς ο κατάλογος. Όλα όλα αυτά χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, γραφειοκρατία, διοικητικές δαπάνε. Υποτίθεται ότι απομακρυνόμασταν από όλα αυτά με την τελευταία μεταρρύθμιση και στην αρχή της μεταρρύθμισης ε, όλοι κάναν ομιλίε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την απλούστευση και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προηγούμενη μεταρρύθμιση. Όμω ε, οπισθοδρομούμε σε σχέση με αυτό και κάτι άλλο που δεν προανέφερε κανένα, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό και ε, λυπάμαι ιδιαίτερα για την απώλεια του στόχου και της δεδηλωμένης πρόθεσης του Κοινοβουλίου να επικρατήσει πλήρης διαφάνεια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό ζήτησε το Κοινοβούλιο και εξέλιψε τελείως. Είναι θλιβερό. Γέγγλε και Σικερέσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα θυμάστε σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει πόσο μεγάλη απόκληση παρουσιάζαν οι θέσεις μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, ιδιαίτερα εσάς, για τα βήματα προσέγγισης που κάνατε και εσάς κύριε Προεδρεύον Ιδιαιτέρως που ακούσατε και παρακολούθησατε τις θέσεις των προσώπων των πολιτικών ομάδων, των συντονιστών. Βεβαίως Ξέρω πόσο δύσκολη ήταν η διαπραγμάτευση. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Μισελ Ντοντά. Ξέρω ότι δεν συμφωνεί η γερμανική κυβέρνηση σε όλα τα σημεία. Μπορούμε να το προβλέψουμε άλλωστε αυτό. Θεωρώ ωστόσο ότι η συμφωνία στην οποία καταλήγουμε μας επιτρέπει και να μεριμνήσουμε για την οικονομία και να ενισχύσουμε περισσότερο την οικολογία, που ίσως κάποιοι άλλοι οικολογικοί αυτοί θα ήθελαν να την προβάλλουν περισσότερο, αλλά πάντως και να έχουν μια καλή γεωργική πολιτική. Και η ερώτησή μου και παράκληση είναι δεν λύγει το θέμα με τη σημερινή συζήτηση. Δεν έχουν εξαντληθεί όλες τις πραγματεύσεις, δεν ψηφίζουμε οριστικά, αλλά μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο με ασφάλεια για όλους τους γεωργούς, για όλους εκείνους που εξαρτάται από το πολιτισμό στο νομικό πλαίσιο τελευταία ανάλυση, για το μέλλον, για να μπορούν να προβλέπουν τα περαιτέρω βήματα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πάνω στο οποίο να μπορούμε να στηριχτούμε για να καταλήξουμε σύντομα σε καλά αποτελέσματα. Συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελίζα Μπεθ, Σικυρέσκη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να διαισθανθούμε ένα γενικό κλίμα αισιοδοξία εδώ σε αυτή την αίθουσα. Γιατί και επιτύχαμε αρκετά και ε, φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε ακόμα ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε και έχουμε όλοι κουραστεί άλλωστε. Ε, βέβαια ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι θέμα του Κοινοβουλίου ούτε, ε, του, ε, ούτε της Κομισιόν. Το Συμβούλιο έχει επιβάλει αυτό το μείον 11% και επομένως πολλοί ήταν αυτοί οι στόχοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν. Αύξηση των άμεσων πληρωμών, και μάλιστα στο δεύτερο πυλώνα μερικές χώρες ε, έχουν μείωση μέχρι και 30% των πληρωμών. Ε, μπορούμε βέβαια να πούμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έχουμε κρίση, αλλά γενικά ενισχύσαμε την θέση των, ε, των γεωργών στην αγορά μειώσαμε τις ενισχύσεις αλλά προτείνουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του γεωργού στην οργάνωση της αγοράς. Προτείνουμε νέους ε, ρυθμιστικούς μηχανισμούς όσον αφορά ε, τα στοιχεία τα οποία συνδέονται με την κρίση. Πολύ σημαντικό στοιχείο ε, και πρέπει εδώ να δείξουμε μεγάλη συνοχή Επίση στηρίξαμε, ε, δεν μπορώ να πω ότι στηρίξαμε τρομερά την, ε, τα έσοδα των γεωργών, αλλά ε, η ΚΑΠ πλέον έχει γίνει και περιβαλλοντική πολιτική, γι' αυτό πρέπει να το πούμε σαφώς. Δύο πράγματα τέλος. Πρώτα απ' όλα να μην λησμονούμε ότι οι περιοχές υπαίθρου θα πρέπει ε, να καλύπτονται και από την πολιτική συνοχή, η οποία μέχρι τώρα υπερβολικά έχει επικεντρωθεί στις αστικές περιοχές και επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει και σύγκληση προς τα έξω. Θα πρέπει οι αγορές να είναι πιο εξωστρεφείς. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της ε, ε, ΚΑΠ άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς προς τα έξω, γιατί έτσι πραγματικά θα έχουμε μια καλύτερη ολοκλήρωση. Επομένως όλες αυτές ε, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι σαφείς. Highland και μετά Αντιπρόεδρος Πότς. Όπως και προλαλήσατε, ε, θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους ε, της διαπραγματευτικής ομάδας, διότι εργάστηκαν σκληρά και για πάρα πολύ καιρό, κυρίως τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα όλος ιδιαίτερος να συγχαρώ τον Υπουργό και την ομάδα του ήταν πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες ε, και επεξεργάστηκαν σωστά τους φακέλους. Ε, ξέρουμε ότι είμαστε σε απάτητο έδαφος μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά όλοι έδωσαν τον καλύτερο ε, εαυτό τους. Σε σχέση τώρα με το ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου βάσει της νέας ε, δομής για τη συναπόφαση, θα πρέπει να αντλήσουμε τα δέγματα του παρελθόν και να κάνουμε τις απαιτούμενε αλλαγές. Ήδη μιλήσαμε για 8.000 τροπολογίες που έπρεπε να περιμένουμε, σύν τις τροπολογίες ολομέλειας και ατελείωτες ώρες ψηφοφορίας. The question of manpower already... Ε, και θα ήθελα τώρα να σας πω για την διαπραγματευτική ομάδα του ε, Συμβουλίου ότι πρέπει να θυμηθούμε ότι ε, το καλύτερο θα ήταν οι εκπρόσωποι των τριών θεσμικών οργάνων να καταφέρουν να συνεννοηθούν γιατί θα ανακύψουν πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον ακόμη και με αυτές ε, τις μεταρρυθμίσεις. Ε, ε, δεν είναι απολύτως απαράδεκτο τα χρηματοοικονομικά ζητήματα να μένουν εκτός διαπραγματεύσεων και να θεωρούνται ως ιερά. σε σχέση με τη διαδικασία θα ήθελα να τονίσω ότι είναι αδύνατο να εκπροσωπήσουμε πλήρως και αποτελεσματικά τα συμφέροντα των γεωργών όταν μας δίνουν τελευταία στιγμή βασικές πληροφορίες. Ε, έχουμε ηθική υποχρέωση και καθήκον ενώπιον των γεωργών να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ε, και όχι να λαμβάνουν άλλοι αποφάσεις ε, εξ ονόματός τους. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομος, κάνω όμως κάποια γενικά σχόλια. Καλωσορίζω την ευελιξία που κατοχυρώθηκε για τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος τους τώρα είναι να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν σωστά αυτά που αποφασίστηκαν. Ε, νομίζω όμως ότι σε σχέση με όλα αυτά που συνέβησαν, οι εξελίξεις είναι θετικές ε, για τους γεωργούς. Ε, οι λιγότερο ευνοούμενες περιοχές, το έλεγα αυτό ανέκαθεν, είναι άλλο σημαντικό πρόβλημα, εξαιρετικά περιπλοκό. Παρόλα αυτά, λήφθη η απόφαση και κάποιοι καλωσόρισαν τα ισχυρά μέτρα υπέρ των νέων γεωργών. Ας σκεφτούμε όμως ότι αυτή είναι και η πιο καινοτόμα πρόταση του μεταρρυθμιστικού πακέτου. Τέλος, ε, θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις σε σχέση με το τι εννοούμε εξισορρόπηση της αγοράς ή διόρθωση των ανισορροπιών. Ε, παραδείγματος χάρη για τις θυλάζουσες αγελάδες ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ιρλανδία να γίνουν απαιτούμενες αλλαγές ε, και οι παραγωγικοί γεωργοί που έκαναν που επέτυχαν τα αποτελέσματα ε, της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ανταμυφθούν. Ε, Υπουργέ ε, θα πρέπει να επιμείνουμε στην απλούστευση και τη μείωση της γραφειοκρατίας ε, διότι είναι ο ακρογωνιαίος ελίθος του όλου εγχειρήματος ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυρία Πόλσεν και μετά ο Λρίκε Ρόντουστ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν και κυρίως τους υπαλλήλου της Γραμματείας. Εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Όλοι εργάστηκαν πάρα πολύ καλά και το κλίμα των διαπραγματεύσεων ε, κυρίως στο τμήμα της Υπέθρου όπου εργάστηκα και εγώ χαρακτηρίστηκε από ένα εξαιρετικά επικοδομητικό πνεύμα και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ε, όμως δεν αρκεί να επιχαίρουμε για την καλή δουλειά που κάναμε, διότι υπάρχει μία λεπτομέρεια ε, την οποία θα έπρεπε να πάρουμε στα σοβαρά όλοι μας. Ε, πώς μπορούμε όλοι να σιωπούμε πούμε για αυτό ε, για το οποίο δεν έχουμε προφανώς δικαίωμα να διαπραγματευόμαστε παρά την ύπαρξη της συνθήκης της Λισαβόνας οι κρατών και κυβερνήσεων και κλεισμένων των θυρών ε, και ε, ε παίρνουν τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό. Δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ εφόσον έχουμε τη Δημοσιονομική Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνούμε να σιωπούμε όλοι και να δεχόμαστε φοβόμαστε ε, ότι δεν συζητείτε τίποτα για τον προϋπολογισμό και να θεωρείτε αυτό ως λεπτομέρεια. Μα πώς είναι δυνατόν. Όλα είναι διαπραγματεύσιμα. Ε, δεν μιλάω για την κοινή γεωργική πολιτική. Εγώ μιλώ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών και έλλειψη, δημοκρατικό έλλειμμα σε αυτό το σύστημα που έχουμε καθιδρύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι όντω το Κοινοβούλιο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά παρότι είχε επικρατήσει ένα συνολικό χάος στην απαρχή της διαδικασίας όλα αυτά τα καταφέραμε. Ευχαριστώ. Ούλρικ ε, Ρόντοστ. Κυρία Ρόντοστ, θα ήθελα να ευχαριστώ την ομάδα διαπραγμάτευσης. Είναι μια μάχη του Γολιάθ κατά του Δαβίδ, όχι καλύτερα του Δαβίδ κατά του Γολιάθ πρέπει να πω και έχει αποδειχθεί ότι ο Δαβίδ πάντα κερδίζει. Γιατί αν κοιτάξουμε τι είδους διοικητικό μηχανισμό είχε πίσω τη σημεία πλευρά και τι είδου είχαμε εμείς με τους λίγους ε, γραμματεί και προσωπικό. Ε, για κοιτάξτε, τουλάχιστον δείξτε και λίγο σεβασμό και αναγνώριση. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια νέα μεταρρύθμιση στην αρχή αυτής της, ε, της πρωτοβουλίας εγώ περίμενα ότι θα μιλούσαμε για πρασίνισμα, κοινωνική διάσταση στη γεωργία, ανταγωνιστικότητα στη γεωργία, σεβασμό από τον πολίτη για τη γεωργία. Αυτό δε και για την οικολογική αλλά και για την παραδοσιακή, για την συμβατική καλλιέργεια. Θέλουμε μέσα, θέλουμε τρόφιμα φθηνά οικονομικά, καθαρά όμως και υγιεινά για τον ε, πολίτη και λιγότερη γραφειοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθεί η λύση και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πρέπει και ο Γεωργός και η διοίκηση να γνωρίζει σύντομα μέχρι, πόσα, μέχρι τι πόσα μπορούν να περιμένουν. Δεν Πρέπει να επιδεινώσουμε εμείς από πλευρά μας τα πράγματα, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια είναι η κατανομή των ποσών, ποια είναι η συγχρηματοδότηση, τι είδους ε, μεταφορά, ε, μεταφορά ποσών θα έχουμε από την πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Και εκ είναι πολύ δύσκολο με βάση τα στοιχεία που έχω στη θέσή μου να αποδεκτώ αυτό ε, που βλέπω ως τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με την αρχική μου ε, προσδοκία. Εάν δεν δεχθεί λοιπόν το στο δημοσιονομικό πλαίσιο του Συμβούλου, τα πράγματα δεν θα είναι πιο εύκολα στο μέλλον. Και ενδέχεται να συνεχίσουμε να μαρτυρόμαστε και να φτάσουμε και μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν λοιπόν δεν δοθεί σύντομα μία λύση, μπορούμε να καταλήξουμε ακόμα και στην απόρριψη της προτάσεως. Θέλουμε μία γεωργία αποτελεσματική, λειτουργική, ανταγωνισματική. Σε κάποιους τομείς το έχουμε καταφέρει, σε κάποιους όχι. Η πολιτική όμως είναι η τέχνη των συμβασμών και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αν πράγματι επιτύχαμε στο βαθμό που μπορούμε να δεχθούμε λύσεις. Θα πρέπει να συνομιλήσω βεβαίω με την ομάδα μου, τη Σοσιαλιστική Γερμανική Αντιπροσωπεία. Έχουμε όμως ανοίξει έναν δρόμο για, την, για το πρασίνισμα της γεωργίας, για την πιο οικολογική γεωργία και μπορούμε χάρη σε αυτήν να δώσουμε λύσεις και για τους γεωργούς. Θα έχουμε σε μερικά χρόνια πάλι μεταρρύθμιση ίσως και γι' αυτό ελπίζω να μην σκεφτεί κανείς, να μην διανοηθεί κανείς να κλείσει αυτή την ανοιχτή πόρτα. Ευχαριστώ πολύ, ο Αντιπρόεδρος Panie Przewodniczący, e, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως, η εργασία που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη και το τελικό έγγραφο είναι πολύ καλύτερο από το αρχικό. Μπορέσαμε δηλαδή να βελτιώσουμε πολλές ε, προτάσεις ε, της ε, Κομισιόν και επομένως αναγνωρίζω την προσπάθεια και του Προέδρου και των εισηγητών και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια η εργασία είναι θετική. Όμως πρέπει να αναφερθώ και στις ανησυχίες μας. Μη λησμονούμε ότι ολοκληρώνουμε τις εργασίες αυτές για την ΚΑΠ μια ΚΑΠ η οποία όμως εξακολουθεί να είναι πολιτική διακρίσεων και διακριτικής μεταχείρισης. Ήδη στην ΚΑΠ μιλάμε για ε, παλαιά και νέα μέλη. Ε, ε, χώρες οι οποίες ε, παίρνουν περισσότερα και άλλες που παίρνουν λιγότερα. Δηλαδή τι, οι πλούσιοι παίρνουν περισσότερα και οι φτωχοί παίρνουν ακόμα λιγότερα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Εγώ εδώ πρέπει να ασκήσω κριτική. Πρόκειται για διακριτική μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διακρίσεις και όσο και αν προσπαθούμε να αμβλύνουμε την εικόνα αυτή είναι εδώ και υπάρχει. Άλλο σημείο η πολιτική προστασία του περιβάλλοντος. Και εδώ υπάρχει κάποια υποκρισία. Ε, εξαίρετη ιδέα είναι αυτό το πρασίνισμα, το greening, αλλά εδώ θέλουμε πραγματικά να προστατέψουμε το περιβάλλον ή μήπως θέλουμε να παράγουμε λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εισάγουμε περισσότερα από τα παραγόμενα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, προϊόντα. Θέλουμε πραγματικά να, μειώσουμε, να, να βελτιώσουμε την παραγωγή ή θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι κάποιων βιομηχάνων. Τι θα γίνει, θα, μήπως πρέπει να βγάλουμε απ' έξω τις μεγάλες, ε, ε μεγάλες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, οι οποίες πολύ κακό κάνουν στη, στο περιβάλλον. Τώρα στρέφομαι και προς τον πρόεδρο Δεκάστρο γιατί και η Πολωνία όπως και η χώρα του έχουν περίπου το ίδιο πρόβλημα όσον αφορά δηλαδή τα προϊόντα, την παραγωγή προϊόντων καπνού. Τι θα πρέπει να πω εγώ σε 15.000 ανθρώπους, θα τους πω δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ε, να πάτε κάπου αλλού, να, τι να σας πω, να πάτε στην Ιρλανδία ας πούμε και να σας βρει δουλειά η κυρία Μαγκίνες. Ε, θα πρέπει να φύγετε από τη χώρα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. 15.000 άνθρωποι οι οποίοι χωρίς επιδοτήσεις δεν θα μπορέσουν να ε, ξεπεράσουν και τα προβλήματά τους και να επιβιώσουν. Δεν ξέρω αν και στην Ιταλία το πρόβλημα είναι ίδιο. Πάντως σε εμά οι παραγωγοί καπνού έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και λυπούμε ειλικρινά που δεν επετεύχθη ε, συμφωνία, συμφωνία στα πλαίσια του Συμβουλίου. Και εδώ έχουμε επομένως πολιτική ε, διάκριση. Γι' αυτό ήθελα εγώ να πάρω τον ε, λόγο, ε, γιατί αυτή η διακριτική μεταχείριση σκιάζει λίγο τη γενικότερη χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ Σαρβάνα και μετά Καδινόσκι. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό εγώ θα ασχοληθώ μόνο με το πρασίνισμα, με το greening το greening, το πρασίνισμα ήταν η κεντρική λέξη, η λέξη κλειδί αυτής της μεταρρύθμισης και χαίρομαι ε, που είναι λογική η μεταρρύθμιση γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια ε, βαθυτάτη διαφορά ανάμεσα σε πολιτικές όπως είναι η οικονομική πολιτική, η εφαρμογή και η υλοποίηση της ε, εσωτερικής αγοράς από τη μία και ε, την γεωργική πολιτική από την άλλη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ζητήσουμε τα ίδια, τα, ίδια μέτρα πρασίνισματος ε, από μια χώρα η οποία έχει μόνο ε, χωράφια και το, την ίδια προσπάθεια πρασινίσματος σε μια χώρα που έχει μόνο λίμνες ας πούμε. Χαίρομαι, χαίρομαι που έχουμε το greening και τα όσα από αυτό προβλέπονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σλεύς Καντινόφσκι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σαν γεωργός εγώ ο ίδιος θα επαναλάβω αυτά που είπε ο ε, συνάδελφος Νίκολσον. Με λιγότερα χρήματα πρέπει να κάνουν περισσότερα ε, οι γεωργοί. Λυπούμε κι εγώ, όπως και άλλοι, που δεν θα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τις άμεσες ε, πληρωμές. Και όσον αφορά την εξωτερική σύγκληση, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι ιστορικές αναφορές. Με αυτή την έννοια εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αδικία και μεγάλες διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, μεγαλύτερη νομιμότητα θέλαμε της ε, πολιτικής ε, στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών φορολογουμένων. Ε, ένα 30% του δεύτερου πυλώνα θα δοθεί για το περιβάλλον Τέλος πάντων, τότε να μην ονομάζουμε την πολιτική αυτή ε, ΚΑΠ, να, την ε, μιλά, να μιλάμε για ε, γεωργική και περιβαλλοντική πολιτική. Εκεί θα είμαστε πιο νόμιμοι. Επίσης, 2% για, την, για τις παραγωγές Αλλά νομίζω ότι εδώ δεν μπορούμε να, να διευρύνουμε περισσότερο τις πρωτεϊνικές παραγωγές Ενδεχομένως ε, εδώ θα υπάρξει επικάλυψη ε, και με τα περιβαλλοντικά, ε, με τις περιβαλλοντικές καλλιέργειες. Πρόεδρος. Και abbiamo un sostegno politico ampio all'accordo che abbiamo raggiunto come team negoziale. Πρόεδρος, νομίζω ότι πρέπει να πω ότι εδώ έχουμε μια ευρεία συμφωνία. Μας ικανοποιεί πάρα πολύ ε, και τους εισηγητές ε, και τους εισηγητές και την Προεδρία και την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Νομίζω ότι μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι η πολιτική συμφωνία ε, στηρίζεται από τους περισσότερους. Βεβαίως ευελπιστούμε πλέον ότι οι διαπραγματεύσεις για τις πιδέλταπή για το πει και τις δημοσιονομικές προοπτικές θα ολοκληρωθούν. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους και νομίζω ότι μπορούμε ε, να ολοκληρώσουμε αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Γεωργίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους παριστάμενους. Ε, βλέπω ότι έχουμε εδώ πέραν των συνήθων ε, μελών και ε, τα λοιπά. Βλέπω και εκπροσώπους των γεωργών, βλέπω και πολλούς ενδιαφερόμενους. Ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή μάλλον και σε λίγο στην ίδια αυτή αίθουσα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Ευχαριστώ.